Αγαπητοί συνάδελφοι, ας ξεκινήσουμε τη συνεδρίαση. Ως ε, συνήθως ε, αναμεταδίδεται και από το διαδίκτυο. διαδίκτυο. Περνάμε στο πρώτο θέμα, έγκριση μερίσιας διάταξης. Ε, σχετικά έχω δύο-τρία ενημερωτικά. Πρώτον, υπάρχει ο κύριος Ούγκιας, ο οποίος ενημέρωσε την γραμματεία ότι δεν θα μπορέσει να έρθει σήμερα και άρα η, η συζήτηση για τη γνωμοδότησή του που είναι το υπερθμό 6 προτείνεται να μετακινηθεί στην αυριανή πρωινή συνεδρίαση μετά το 8 την έκθεση του Φρανσουάλ Φοντσί, ε, Στο πλαίσιο αυτό Θέλω να ζητήσω κάποια, ε, το, τον κύριο Αλφόνση να δείξει κάποια ευελιξία. Αν έχουμε σήμερα χρόνο, μπορούμε να το συζητήσουμε σήμερα το δικό σας θέμα και ίσως και να το τελειώσουμε αν έχουμε χρόνο, να μην πιεζόμαστε αύριο. Και κατόπιν, μετά την παρουσίαση μάλλον την ανταλλαγή απόψεων με την κυρία Υπουργό, θα ήθελα να σας ενημερώσω εγώ ε, σύντομα για το τι περιλαμβάνεται στο σημείο 10 της ημερήσιας διάταξης, όπου υπάρχει αυτό το ε, μέσο επιμερισμού του κινδύνου. Θα ήθελα να σας ενημερώσω δεν θέλω να γίνει τώρα συζήτηση, θα σας τα εξηγήσω όλα, αλλά όλα αυτά αφού γίνει η ανταλλαγή απόψεων με την κυρία Υπουργό. Αυτές είναι λοιπόν οι πιθανές αλλαγές τροποποίησης στην ημερήσια διάταξη. Αν δεν έχετε αντίρρηση μπορούμε να την εγκρίνουμε. Και όσον αφορά το σημείο 2 που αφορά την έγκριση των πρακτικών της προηγούμενης έκτακτης συνεδρίασής μας στις 14 Νοεμβρίου, τα πρακτικά έχουν κυκλοφορήσει και θα θεωρηθούν, θεωρηθεί ότι, έχει εγκριθεί, ότι έχουν εγκριθεί ως συνήθως αν μέχρι το τέλος της συνεδρίασης δεν έχει κάποιος θέσει θέμα για τις ανακοινώσεις Πρόεδρου. Όπως ήδη σας είπα, θα κάνω τις ανακοινώσεις μου μετά την ανταλλαγή απόψεων που θα έχουμε με την κυρία Ελσβιέτα Μπινκόφσκα που είναι Υπουργός Περιφερειακής Ανάπτυξης ε, της ε, Πολωνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η οποία θα μιλήσει για θέματα που αφορούν εμάς, την πολιτική συνοχής. Η Προεδρία ολοκληρώνεται, ο χρόνος ε, περνάει πάρα πολύ γρήγορα. Την προηγούμενη εβδομάδα έγινε το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων που ασχολήθηκε ακριβώς με αυτή την πολιτική και είμαι βεβαία ότι όλα αυτά θα θέλει να μας τα πει η κυρία Υπουργό και μετά θα ακολουθήσει η συζήτηση. Χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση λοιπόν θα δώσω το λόγο στην Υπουργό της Πολωνίας, την κυρία Μπινκόφσκα να πάρει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Πραγματικά ο χρόνος ε, περνάει ταχύτατα. Θυμάμαι πολύ καλά όταν συναντηθήκαμε στις 2 Ιουλίου για πρώτη φορά στο πλαίσιο της ε, Πολωνικής Προεδρίας στο Συμβούλιο Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Περιφερειακή Ανάπτυξη και τώρα ολοκληρώνεται η Προεδρία. η στιγμή της Πολωνικής Προεδρίας έγινε σε μια πολύ ιδιαίτερη στιγμή της Ευρωπαϊκής, ε, των ευρωπαϊκών θεμάτων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Ιούνιο παρουσίασε την ανακοίνωση του προπολογισμού για την περίοδο 2014-2020 και αργότερα τον Οκτώβριο τα νομοθετικά πακέτα για κάθε μια από τις πολιτικές. Και έτσι ξεκίνησε η επίσημη συζήτηση για το τι θα γίνει σε κάθε μια από αυτές τις πολιτικές και το πώς αυτές θα εφαρμοστούν. Ταυτόχρονα, αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μια οικονομική κατάσταση πολύ καλά γνωστή σε όλους μας. Η συζήτηση αυτή ήταν εξαιρετικά δύσκολη κάποιες στιγμές, παρότι προσπαθήσαμε να προσαρμόσουμε το ρυθμό και στο χρονοδιάγραμμα που σας παρουσίασε τον Ιούλιο, προσπαθήσαμε να το τηρήσουμε. Στα διάρκεια της πολιτικής Προεδρίας η πολιτική συνοχής είναι μια συγκεκριμένη και πολύμορφη ανταπόκριση στις ανάγκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η βασική στόχη που είχαμε θέσει ήταν η ενίσχυση όλων των χαρακτηριστικών της πολιτικής αυτής μέσω μιας ολοκληρωμένης και ε, επικεντρωμένης ε, χωροταξικά προσέγγισης. Σχεδόν όλα όσα συζητήσαμε ε, ε, αφορούσαν αποτελέσματα. Είχαμε συμφωνήσει ότι θα επικεντρωθούμε σε αποτελέσματα. Η συζήτηση Στη συζήτηση κυριάρχησε τα θέματα της Επιτροπής 13 του Συμβουλίου, την ομάδα εργασίας ε, για τα διαρθρωτικά ταμεία. Εκεί ε, τα κράτη-μέλη παρουσίαζαν τις αρχικές απόψεις, ε, οι στάσεις τους για τη θεματική συγκέντρωση, τη και τα μέσα για την χωροταξική ανάπτυξη. Τις λεπτομέρειες θα τις παρουσιάσω αργότερα. Θεωρώ όμως ότι ο στρατηγικός προγραμματισμός και η επικέντρωση σε κάποια θέματα είναι χώροι τομείς στους οποίους σημειώθηκε σημαντική πρόοδος. Και τώρα θα παραδώσουμε στην Δανέζικη Προεδρία ε, μια αρκετά προχωρημένη φάση των θεμάτων αυτών. Οργανώσαμε και τεχνικές συνεδριάσεις για τα ίδια θέματα όπου συμμετείχαν και μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων που θα σας παρουσιάσω σε λίγο, ε, ε, έγινε συζήτηση για την έκθεση, την εργασία του Συμβουλίου και τα επιλεγμένα θέματα που χρειάστηκε να έχουν πολιτική υποστήριξη συζητήθηκαν στο επίπεδο των Υπουργών Υπεύθυνων για την Πολιτική Συνοχή στη διάρκεια του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων. Ε, μια τέτοια συνεδρίαση έγινε πριν από δύο-τρεις μέρες της, ε, την Παρασκευή στις 16 Δεκεμβρίου. Τα κράτη-μέλη θεώρησαν ευπρόσδεκτες τις νέες τάσεις για τις αλλαγές που πρότεινε η Κομισιόν, κυρίως όσες αφορούν την ε, στενή σχέση μεταξύ την ε, πολιτική συνοχής και την Ευρώπη του 2020 πιο ε, μεγαλύτερη ε, προσοχή στην ανάπτυξη και βεβαίως κινήσεις στο τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Όλοι δεχόμαστε ότι όλα αυτά αποτελούν σωστή βάση για διαπραγμάτευση, αλλά όλες οι χώρες γνωρίζουν ότι όλα αυτά πρέπει να συζητηθούν σε ε, βάθος, κυρίως τα μέσα που αφορούν την εφαρμογή της πολιτικής. τα βασικά συμπεράσματα είναι τα εξής. Τα κράτη-μέλη που αποδέχονται τις προτάσεις της Επιτροπής το κοινό στρατηγικό πλαίσιο Όλοι θεωρούν ότι ένα τέτοιο έγγραφο για το στρατηγικό πλαίσιο θα βελτιώσει τη συνοχή τη συνεκτικότητα μεταξύ των εθνικών πολιτικών, των ευρωπαϊκών πολιτικών και της στρατηγικής του 2020. Όμως θεωρήθηκε ότι ο τρόπος με τον οποίο προσεγγίζει η Κομισιόν το θέμα δεν είναι παρικής. Ο τρόπος ε, ε, έγκρισης των προτάσεων ή ε, Κομισιόν πρότεινε κατεξουσιοδότηση πράξη που εγκρίνονται μόνο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έγινε συζήτηση και η Προεδρία πρότεινε το κοινό, το κοινό στρατηγικό πλαίσιο να προταθεί υπό τη μορφή νομοθετικού ψηφίσματος ως παράρτημα δηλαδή του γενικού κανονισμού που εγκρίνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Η λύση αυτή, κατά την άποψή μας, ε, δίνει μεγαλύτερη πολιτική, πολιτικό βάρος αυτό το έγγραφο στην προγραμματική αυτή περίοδο. Η πρόταση αποτελεί κομμάτι το μέρος της φιλοδοξίας που έχει η Πολωνία να ενισχυθεί η σημασία της ε, πολιτική συνοχή στη γενικότερη αρχιτεκτονική των ευρωπαϊκών πολιτικών. Πρέπει να σας πω ήδη ότι έγινε θετικά δεκτή αυτή η πρόταση. Όλες οι χώρες μέλη πλην μιας ε, που είχε κάποιους δισταγμούς κατά την επίσημη συνάντηση των Υπουργών στις 16 Δεκεμβρίου. Δεύτερον, πρέπει να βελτιωθεί η συνοχή μεταξύ εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών όπως σας είπα και ανάμεσα στην, και στην ε, στρατηγική Ευρώπης 2020. Γι' αυτό τα περισσότερα κράτη-μέλη διατύπωσαν αμφιβολίες και ερωτήματα σε σχέση με τις ε, προτάσεις κομισιών για τους μηχανισμούς και τις ε, προτάσεις, τις συστάσεις που γίνονται σε κάθε χώρα κατέτος που αποτελούν σημείο αναφοράς για την επιλογή των θεματικών στόχων. Στη διάρκεια της επίσημης συνάντησής τους οι Υπουργοί αντιτάχθηκαν όλοι σε αυτή την προσέγγιση ε, είπαν ότι αυτού του είδους τα, το έγγραφο δεν είναι το πλέον κατάλληλο και ότι πρέπει να δούμε ποιες θα είναι οι μεταρρυθμίσεις που γίνονται. Τα κράτη-μέλη θεωρούν ότι οι συμβάσεις εταιρικής σχέσης ε, και σε κοινοτικό επίπεδο θα έπρεπε να αποτελούν το γενικό πλαίσιο του προγραμματισμού. Τα κράτη-μέλη υπογράμμισαν με έμφαση ότι θα πρέπει να εξορθολογιστεί το, το περιεχόμενο των προγράμματων και των συμβάσεων, να μην υπάρξουν αλληλεπικαλύψεις και βεβαίως να μελετηθεί η σκοπιμότητα. Η Κομισιόν τώρα μελετά ένα νέο θέμα, επί του οποίου θα επανέλθω, πρόκειται για μια πρόταση που στόχο έχει τη δημιουργία ενός νέου μηχανισμού ε, που θα συγκεντρώνεται σε συγκεκριμένα θέματα, το λεγόμενο ring fencing. Τα κράτη-μέλη τώρα από πλευρά του είναι υπέρ ε, αυτής της συγκέντρωσης των πόρων ε, για, τα, για τους μεγάλους άξονες, όμως ταυτόχρονα θέλουν όλοι να επισύρουν την προσοχή στο γεγονός ότι θα πρέπει εδώ να υπάρξουν και προϋποθέσεις ε, όροι για τις περιφέρειες, για τα κράτη κλπ. Και αυτό παρουσιάστηκε και ε, ως θέμα στο Συμβούλιο της 16ης Δεκεμβρίου. Η Προεδρία πρότεινε να ξανασυζητηθούν τα θέματα αυτά όταν θα γίνουν οι διαπραγματεύσεις. Δεν θα πρέπει δηλαδή να επιβάλλονται όλα αυτά. Τα κράτη-μέλη είναι υπέρ της πολλαπλής συμμόρφωσης, δηλαδή πρέπει να υπάρχουν τις ε, της αιρεσιμότητας για να μην υπάρχει πρόβλημα, γιατί χωρίς αυτό δεν υπάρχει σωστή απεικόνηση πραγματικότητας. Πολλοί φόβοι αναφέρθηκαν για αυτή την αιρεσιμότητα την μακροοικονομική αιρεσιμότητα η οποία ξεπερνά τα πλαίσια της πολιτικής συνοχής και της αρμοδιότητας των κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τα κράτη-μέλη ε, είχαν θετική στάση ε, για την ενίσχυση των μέσων της ε, το, της, χωροταξ... της περιφερειακής ανάπτυξης. Υπάρχουν ε, ένας πολλαπλασιασμός των μέσων για το ΦΕΝΤΕΡ και λοιπά, αλλά εδώ το σύστημα περιπλέκεται, δεν απλουστεύεται όπως επιθυμούμε. Όπως σας είπα, η Πολωνική Προεδρία κατάφερε να προχωρήσει σημαντικά σε δύο χώρους. Το στρατηγικό προγραμματισμό και την ε, συγκέντρωση των θεμάτων. Υπάρχει και το θέμα της αιρεσιμότητας και το θέμα της ε, του χωροταξικού σχεδιασμού. Επανειλημμένος ε, στο πλαίσιο του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων έγινε συζήτηση για αυτά τα θέματα, πράγμα που αποτελεί επιτυχία και πιστεύουμε ότι τα πράγματα πρέπει να συνεχιστούν έτσι και ελπίζουμε θα πάνε καλά και σε επόμενες προεδρίες. Υπάρχει κάτι πολύ σημαντικό που καταφέραμε, διαπραγματευτήκαμε τον Γενικό Κανονισμό ε, 1083 Πρόκειται για μέσα, για τη χρηματοοικονομικά και δεύτερον για προσωρινή συγχρηματοδότηση των κρατών μελών που βρίσκονται σε δημοσιονομικά δύσκολη θέση. Και ήθελα να ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που επέδειξε πνεύμα συνεργασίας, αφοσίωση. Σας ευχαριστώ που μπορέσατε να κινηθείτε γρήγορα στα θέματα αυτά. Ως Προεδρία μπορέσαμε να οριστικοποιήσουμε τα, συμπεράσματα των κρατών μελών για όσον αφορά τις συστάσεις για την υλοποίηση της Στρατηγικής Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περιφέρεια της Βαλτικής. Η τελευταία εκδοχή των συμπερασμάτων εγκρίθηκε στην συνεδρία του Συμβουλίου ε, Γενικών Υποθέσεων στις 15 Νοεμβρίου. Επίσης οργανώσαμε ένα ε, σύνολο συνεδριάσεων και συναντήσεων ε, στα πλαίσια της άτυπης συζήτησης. Μιλήσαμε για τα μέσα και τους μηχανισμούς που θα επιτρέψουν την ενίσχυση της ολοκληρωμένης και εδαφικής προσέγγισης για την, τις Πολιτική συνοχή και βεβαίω ε, χρειαζόμαστε αποτελέσματα. Υπήρξε ενεργό συμμετοχή και από πλευρός ε, κράτη-μέλη, από τα θεσμικά όργανα, από τα πανεπιστήμια, του εμπειρογνώμονε και από αυτού που εργάζονται στο πεδίο. Με την ευκαιρία αυτή θα ήθελα να ευχαριστήσω του εκπροσώπου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου γιατί δεν νομίζω ότι υπήρξε ούτε μια συνεδρία στην οποία να μην παρευρίσκεται ε, κάποιο από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Επίσης θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι στην ε, Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης στις 16 ε, και 17 Οκτωβρίου επισκεφτήκατε την Πολωνία. Θέλω να σας ευχαριστήσω για τη δουλειά που κάνατε για το νομοθετικό πακέτο και για το μέλλον, τη συζήτηση που κάνατε για το μέλλον της πολιτικής συνοχής τα πιο σημαντικά συμπεράσματα στα οποία μπορούμε να καταλήξουμε από τις εργασίες του τελευταίου εξαμήνου στην άτυπη αυτή συζήτηση συγκεντρώθηκαν στο πλαίσιο των συμπερασμάτων της Προεδρίας για την εδαφική ε, και πολιτική της και πολιτική συνοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχει και ένα άλλο έγγραφο, δικός χάρτης για την προώθηση και ενίσχυση μιας ολοκληρωμένης και ε, εδαφικής προσέγγισης για να ενισχυθεί η εδαφική ε, ατζέντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το έγγραφο αυτό ε, αποτέλεσε ε, αντικείμενο εκτεταμένης διαβούλευσης με τα κράτη-μέλη, με τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης μεταξύ άλλων και κατά την άτυπη συνάντηση των Υπουργών στις 24 και 25 Νοεμβρίου. Τα συμπεράσματα της Προεδρίας και αυτός ο δικός χάρτης που μόλις ανέφερα δείχνουν ξεκάθαρα ότι υπάρχει σαφή σχέση ανάμεσα στην εδαφικότητα και στην αποτελεσματικότητα. Η αποτελεσματικότητα πρέπει να αποτελέσει βασικό κριτήριο το οποίο να χρησιμοποιούμε για την εδαφική μας προσέγγιση και ε, θα είναι και το, πρέπει να είναι και το τελικό αποτέλεσμα των εργασιών μας. Δεν υπάρχει μία και μοναδική λύση, μία λύση που να μπορεί να εφαρμοστεί παντού σε όλες τις περιοχές και γι' αυτό πρέπει ο προγραμματισμός, οι πολιτικές δράσεις να είναι ευέλικτες και πρέπει να φροντίσουμε οι αποφάσεις να λαμβάνονται στο κατάλληλο επίπεδο για κάθε περιφέρεια. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό η εδαφική προσέγγιση μπορεί να αποτελέσει σημαντικό μέσο για την επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι ε, μέσω αυτής ε, συνδέουμε τις εξωτερικές δράσεις με το ξεχωριστό δυναμικό κάθε περιοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η συνθήκη της Λισαβόνας αλλά και όλες οι εργασίες που έχουν τώρα, μέχρι τώρα πραγματοποιηθεί, ας πούμε η, γραφική ατζέντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2020 μπορούν να αποτελέσουν βάση για αυτή την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο μέλλον. Το σημείο αυτό έχει άμεση σχέση με την ε, ενίσχυση της δράσης στο τοπικό επίπεδο. Πρέπει να γνωρίζουμε ότι οι Δήμοι παίζουν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο, αποτελούν την κινητήρια δύναμη για την ανάπτυξη και είναι κλειδί στην εδαφική ε, ανάπτυξη. Γι' αυτό πρέπει να χρησιμοποιήσουμε μέσα που θα μας επιτρέψουν να λάβουμε υπόψη τις, ε, τα ειδικά χαρακτηριστικά των πόλεων. Ένα άλλο ε, σημείο που θέσαμε είναι η συνεργασία μεταξύ των ευρωπαϊκών περιφερειών. Ε, ε, έχουμε κάνει ένα σχέδιο για το πρόγραμμα της διαμεθοριακής συνεργασίας. Επιπλέον η Προεδρία οργάνωσε συζητήσεις μεταξύ κρατών μελών και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το πρόγραμμα διαμεθοριακής συνεργασίας που πραγματοποιείται εκτός συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χαίρομαι γι' αυτό, διότι όλα όσα έχουμε προβλέψει, δηλαδή η καλή συνεργασία με σκοπό το πρόγραμμα που γίνεται εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης να στηρίζεται στις αρχές της πολιτικής συνοχής έχει γίνει δεκτό από παντού. Η συζήτηση ξεκίνησε στη διάρκεια της δικής μας προεδρίας, εξακολουθεί και θέλω να ευχαριστήσω τη Φιλανδία που διοργάνωσε συνάντηση την περασμένη εβδομάδα για την εταιρική σχέση με μια σειρά από χώρες. Είναι η διαδικασία της Βαρσοβίας, το πλαίσιο της οποίας ε, ε, ασχολούμαστε με τα προγράμματα που έχουν ξεκινήσει εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εν κατακλείδη, αυτή η άτυπη συζήτηση που έγινε το εξάμεινο αυτό ε, έδειξε, έδειξε ότι από πλευράς κρατών μελών υπάρχει ισχυρή θέληση να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα της πολιτικής συνοχής τόσο μέσω ενός ενισχυμένου συντονισμού των, των τομεακών δράσεων, δηλαδή στο κοινό στρατηγικό πλαίσιο, αλλά και μέσω μιας ε, επικέντρωσης προσοχής ε, σε διάφορους θεματικούς άξονες, μια, ένας ενισχυμένος συντονισμός, ένα, ε, μια περιφερειακή διάσταση που να είναι και αυτή ενισχυμένη, όπως επίσης και μια προσπάθεια αξιολόγησης. Είμαι ε, πεπισμένη ότι αυτή η συζήτηση θα συνεχιστεί και κατά τη διάρκεια της Δανέζικης και της Κυπριακής Προεδρίας. Εν κατακλείδη θέλω να σας ευχαριστήσω για μια ακόμα φορά. Ευχαριστώ όλους τους προσώπους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τον εξαιρετικά δραστήριο τρόπο με τον οποίο συμμετείχατε στη διάρκεια της ε, Πολωνικής Προεδρίας και ελπίζουμε ότι στη διάρκεια των επόμενων Προεδριών θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε και να συνεργαζόμαστε για όλα αυτά τα θέματα. Ελπίζω ότι στις δύο επόμενες προεδρίες θα μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε το θέμα αυτό και τις διαπραγματεύσεις για το νομοθετικό πακέτο. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ την Υπουργό. Η κυρία Στρέτερ ζήτησε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ σημαντικό το έργο θεωρώ, της ε, Πολωνικής Προεδρίας. Η διαδικασία είναι νέα και ενοφανής Ποτέ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν είχε στο παρελθόν συναπόφαση. Οπότε έχει σημασία ο τρόπος με τον οποίο προσεγγίζουν τα δύο θεσμικά όργανα το κείμενο του κανονισμού και ήταν πραγματικά πάρα πολύ πολύτιμη δική σας ενισφορά. Σε σχέση με αυτό θα με διέφερε εμένα, ακριβώς για να μπορέσω να εκτιμήσω με ποιο τρόπο Συνεχίζεται η εργασία στο Συμβούλιο. Θέλω να σας ρωτήσω, τις επαφές και συζητήσεις που είχατε, όχι μόνο για αυτά τα θέματα που μας αναφέρατε, αλλά και στις γενικότερες συζητήσεις που κάνατε εκεί για τον κανονισμό. Μπορείτε να μας πείτε ποια σημεία στο κείμενο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, τα απορρίπτει συλλήβδιν το Συμβούλιο. Και δεν υπάρχει καμία αποδοχή ούτε αναμένεται στο μέλλον. Μπορείτε να μας πείτε τα σημεία που είναι κατηγορηματικά αντίθετο Συμβούλιο για να μπορέσουμε λίγο να προσανατολιστούμε, να καταλάβουμε πώς θα διαμορφώσει τη θέση του το Συμβούλιο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Ντελή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και την εκπρόσωπο της Προεδρίας στην ε, δική μας Επίτροπη, η πολιτική συνοχή θα πρέπει να αντιμετωπίσει πολλές προκλήσεις της οικολογίας, της οικονομικές προκλήσεις και τις κοινωνικές, έτσι ώστε να μην υπάρχουν ανισότητες, εδαφικές ανισότητες. Θα ήθελα να ρωτήσω λοιπόν ποιες είναι οι σχέσεις σας με τα κράτη ως προς έναν προϋπολογισμό που θα είναι στο ύψος των περιστάσεων για να αντιμετωπιστούν αυτές οι προκλήσεις. Μιλήσατε και για μακροαιρεσιμότητα. Εμείς, μάλλον το Κοινοβούλιο, αρνήθηκε κάθε μορφή αιρεσιμότητας που βασίζεται στο Σύμφωνο Σταθερότητας. Όμως η Κομισιόν είναι υπέρμαχος αυτών των μέτρων. Αναφέρει ότι αν ένα κράτος μέλος έχει υπερβολικό έλλειμμα και αν δεν επαναπροσδιορίσει την πολιτική του μέσα σε ένα μήνα, μέσα στα, ε, στα πλαίσια της αντιμετώπισης του δημοσίου χρέους, τότε δεν θα, μάλλον θα ανασταλούν οι πληρωμές. Θα ήθελα πω λοιπόν να ρωτήσω το εξή. Η Πολωνική Προεδρία αναγνωρίζει ότι η πολιτική συνοχής δεν είναι ε, ένα μέσον κύρωση κατά κρατών μελών και δεύτερον, γιατί αυτό αποτελεί πραγματικά κίνδυνο. Αν μπούμε σε αυτή τη λογική, τότε θέτουμε σε κίνδυνο τον προγραμματισμό για τη διαχείριση των πόρων και ταμείων. Δεν μπορεί να υπάρχει δηλαδή χρηστή διαχείριση των προγραμμάτων που βρίσκονται σε μια συγκεκριμένη επικράτεια, δηλαδή ως προς την εδαφική συνοχή. Τι μπορείτε να μας προτείνετε. Η κυρία Ρικάινεν, ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Υπουργό για την εξαιρετική αυτή παρουσίαση θα ήθελα να μιλήσω για την περιφερειακή εδαφική συνεργασία, γιατί είχε ενταχθεί πολύ καλά στην ε, πολωνική ατζέντα. Τι γίνεται ως προς τους κανονισμούς, τις διαπραγματεύσεις ε, για τον κανονισμό, ιδιαίτερα που αφορά την εδαφική συνεργασία Υπάρχουν σημεία τα οποία δεν συζητήθηκαν στο Συμβούλιο. Υπήρχαν συγκρούσεις. Ποια ήταν, ποιες ήταν δικές σας προτεραιότητες. Νομίζω ότι θα μπορούσατε να απαντήσετε σε αυτό το πρώτο κύκλο ερωτήσεων. Ευχαριστώ πολύ. Προς την κυρία Σρέτερ θα ήθελα να απαντήσω το εξής. Μίλησε για τα επόμενα βήματα, τις προτεραιότητες δηλαδή της ε, Προεδρίας της Δανίας. Δεν το είπα ε, εξ αρχής, αλλά θα θέλαμε να προχωρήσουμε προς τα εμπρός έτσι ώστε να προχωρήσουμε σε αυτούς τους ε, τομείς, να είμαστε αρκετά προηγμένοι έτσι ώστε να μπορέσουμε να προγραμματίσουμε την εργασία μας. Γι' αυτό μιλήσαμε για στρατηγικό προγραμματισμό και για την ολοκληρωμένη εδαφική προσέγγιση για την ανάπτυξη. Αυτοί οι δύο τομείς ανατίθενται τώρα στην ε, Προεδρία της Δανίας και μετά από το τελευταίο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων είμαστε σε ένα στάδιο που μπορούμε να πούμε ότι τα κράτη-μέλη συμφώνησαν για κοινέ λύσεις. Τώρα, ένας τομέας ο οποίος θα πρέπει να ολοκληρωθεί, που χρειάζεται περισσότερο, περισσότερη εργασία, αφορά την αιρεσιμότητα και, την, και τα μέσα εδαφικής ανάπτυξης. θα πρέπει να γίνει εκτεταμένη συζήτηση από των θεμάτων αυτών. Η κυρία Σρέτερ επίσης ρώτησε ποια θέματα είναι τα πιο ευαίσθητα. Η μακροαιρεσιμότητα θα ήταν το πρώτο, το κάπινγκ καθώς και τα μέσα υποδομών που συνδέουν τα διάφορα τμήματα της Ευρώπης. Αυτή είναι οι τομείς όπου τα κράτη-μέλη έχουν διαφορετικές ε, προσεγγίσεις και δεν έχουν ληφθεί, δεν έχουν γενικές αποφάσεις. σε σχέση με την πολιτική συνοχής για την αντιμετώπιση της τρέχουσας κρίσης, ε, τονίζαμε πάντα ότι αυτοί οι τομείς κινούνται παράλληλα με τις συζητήσεις που αφορούν το πολιετές χρηματοδοτικό δημοσιονομικό πλαίσιο. Νομίζω ότι τα κράτη-μέλη κατανοούν ότι η Πολωνική Προεδρία θέλει να είναι απόλυτα σαφής. Δηλαδή, θεωρούμε ότι η πολιτική συνοχής αφορά τις επενδύσεις κυρίως. Μέσα στα πλαίσια μιας κρίσης μπορούμε να κινηθούμε προς την σωστή κατεύθυνση ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη βεβαίως και τους όρους εργασίας. Δηλαδή προσανατολιζόμαστε προς την ανάπτυξη και αυτό μπορεί να γίνει μόνο μέσω επενδύσεων. Υπάρχουν τα μέσα και είπατε ότι η αιρεσιμότητα αυτή έχει αποφασιστεί de facto. Όπως είπα πριν, ο σύνδεσμος αυτός της μακροαιρεσιμότητας που αφορά συγκεκριμένους μακροοικονομικούς δείκτες, αυτή η αιτιώδη συνάφη, αυτός ο σύνδεσμος αυτό το interface αποτελεί ε, θέμα συζητήσεων, αυτά τα σημεία διαπαφής δηλαδή. Και η πλειοψηφία των κρατών μελών θεωρεί ότι η σύνδεση αυτών των δύο θεμάτων, η μακροοικονομική πολιτική και η αναπτυξιακή πολιτική θα πρέπει να ιδωθεί ως, όχι ως μια μορφή κύρωσης κατά των κρατών μελών ως προς την χρήση των ταμείων Γι' αυτό πιστεύω ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τα κράτη-μέλη που αντιμετωπίζουν πολύ μεγάλη κρίση. Αυτό δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό. Σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία, εδώ άτυπα ημί, το θέμα αυτό μας απασχόλησε ιδιαίτερα. Και τα βασικά θέματα που αντιμετώπισαν τα κράτη-μέλη αφορούν τη συμπερίληψη αυτών των κεφαλαίων μέσα στα προγράμματα αυτά. Και αυτή η οριοθέτηση, αυτό το ring fencing. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Κομισιόν δεν πρόβαλε αναπτυξιακά προγράμματα που είναι ιδιαίτερα για την ε, μεθοριακή συνεργασία. Επίσης, άλλα κράτη-μέλη ήταν αρνητικά ως προς την μείωση του κατοφλίου, ε, δηλαδή μιλήσαμε για ένα 75%. Αυτά τα κατόφλια είναι, θα ήταν χαμηλότερα σε σχέση με τον στόχο 1 της πολιτικής συνοχής, δηλαδή 85%. Μέσα στα πλαίσια της εδαφικής συνεργασίας λοιπόν θελήσαμε να επιτευχθεί μία συμφωνία ως προς τα ιδιαίτερα αυτά θέματα και μας απασχόλησε ιδιαίτερα ο στόχος 1 της πολιτικής συνοχής. Οργανώσαμε την πρώτη τη διάσκεψη που διοργανώθηκε ποτέ ως προς την οργάνωση αυτού του τομέα. Θελήσαμε αυτά τα προγράμματα να γίνουν πιο ορατά στο ευρύ κοινό. Και αυτό έγινε μέσα στα πλαίσια ανοιχτών ημερών ή μέσω συζητήσεων εργασίας. Δεν βρισκόμαστε ακόμα σε ένα στάδιο που μπορούμε να συναγάγουμε συμπεράσματα, αλλά νομίζω ότι αυτός ο κύκλος συζητήσεων μέσω της διαδικασίας της Βαρσοβίας αφορά προγράμματα που βρίσκονται και πολύ κοντά στα εξωτερικά μας σύνορα. Νομίζω ότι όλα κινούνται προς την σωστή κατεύθυνση. Ευχαριστώ κύριο Σταυρακάκης παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Κυρία Υπουργέ, καταρχήν θα ήθελα να σας ε, συγχαρώ για όλες τις δραστηριότητες και πρωτοβουλίες που έχετε αναπτύξει για την πολιτική συνοχή στο πλαίσιο της Προεδρίας. Ω σημαντικότερη εξ αυτών θα ήθελα να ξεχωρίσω τα συμπεράσματα της Προεδρίας για την εδαφική διάσταση των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη μελλοντική πολιτική συνοχή που παρουσιάστηκαν πρόσφατα στο ε, Πόσναν. Ω Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποστηρίζουμε την ανάγκη συγκέντρωση των επενδύσεων σε ορισμένου στόχου. Δεν πρέπει όμω να παραβλέπουμε το γεγονό ότι οι 11 θεματικοί στόχοι που καθορίζονται από τον Γενικό Κανονισμό σε συνδυασμό με τι ειδικέ προβλέψει των κανονισμών για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακή Ανάπτυξη και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο καταλήγουν να περιορίζουν σημαντικά του τομεί όπου κάποιε περιφέρειες μπορούν να επενδύσουν. Και στο πλαίσιο αυτό δεν πρέπει να υποτιμάμε τον κίνδυνο ενίσχυση μια τομεακή προσέγγιση εκεί όπου στόχο μα θα πρέπει να είναι η ενίσχυση τη ολοκληρωμένη προσέγγιση, κάτι το οποίο έχουμε κατά επανάληψη τονίσει σε πολλά ψηφίσματά μα. Τα συμπεράσματα λοιπόν τη Προεδρία αναδεικνύουν ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα τη πολιτική συνοχή μέχρι τώρα. Και αυτό είναι η ικανότητά τη να προσαρμόζεται στι διαφορετικέ ανάγκε και τα χαρακτηριστικά κάθε περιφέρεια. Η προστιθέμενη της αξία έγκυται ακριβώς σε αυτή την ικανότητα να εντοπίζει τις περιφερειακές προκλήσεις και αναπτυξιακές ευκαιρίες που παρουσιάζει κάθε περιφέρεια και να συμβάλλει στην υλοποίηση ευρωπαϊκών στόχων μέσα από στρατηγικές που βασίζονται στα εδαφικά χαρακτηριστικά της εκάστοτε περιφέρειας. Αυτό υπήρξε ανέκαθεν... Αυτό υπήρξε ανέκαθεν ένα από τα κυριότερα χαρακτηριστικά της πολιτικής συνοχής αλλά αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα με την ενσωμάτιση του στόχου της εδαφικής συνοχής στη συνθήκη της Λισαβόνας, καθώς και με την ανάγκη νομιμοποίησης της συμβολής της πολιτικής συνοχής στην υλοποίηση ευρύτερων στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως είναι αυτή της Ευρώπης 2020. Έχουμε όμως φτάσει σε ένα σημείο όπου οι στόχοι της πολιτικής συνοχής για την επόμενη περίοδο έχουν ως σημείο αναφοράς και καθορίζονται από την Ευρώπη 2020 και ταυτόχρονα έχουμε αφήσει κατά μέρο ένα από τους βασικούς και κατοχυρωμένους από τις συνθήκη στόχους της πολιτικής συνοχής. Στην πρόταση της Επιτροπής, ο στόχος για εδαφική συνοχή φαίνεται να περιθυροποιείται από τους θεματικούς στόχους της Ευρώπης 2020. Καλωσορίζω λοιπόν τα συμπεράσματα της Προεδρίας σε αυτόν τον τομέα. Ως Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να κατοχυρώσουμε ότι όλοι οι κανονισμοί που θα εγκρίνουμε θα υπηρετούν σε συγκεκριμένους τρόπους και ξεκάθαρα το στόχο της Εθνικής Συνοχής. Ευχαριστώ. I understand there was no really no question but, but comments, but if Εξ όσων αντιλαμβάνομαι δεν υπήρξε ερώτηση, αλλά αν θέλει κυρία Υπουργό να σχολιάσει, ευχαριστώ. Ε, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρο, θέλω και εγώ όπως και οι προλαλήσαντες να ευχαριστήσω την Πολωνική Προεδρία που έδωσε έμφαση στην περιφερειακή πολιτική. Ε, ξέρω ότι είναι δύσκολο ε, για εσά στη φάση αυτή να μα πείτε ακριβώ ποια πρόκειται να είναι η άποψη του Συμβουλίου, γιατί τα κράτη-μέλη έχουν διστάμενε απόψει για το μέλλον τη ε, πολιτική συνοχή. Είναι σημαντικό ω Επιτροπή σήμερα εδώ, δεδομένου ότι σα έχουμε να πάρουμε όσο το περισσότερες απαντήσεις. Υπάρχει ένα θέμα της μακροαιρεσιμότητας, το καλύψατε, όμως είναι και άλλα θέματα που θα ήθελα να ανακαλύψετε. Το θέμα του, ε, του, ε, του αποθεματικού επιδο, ε, επιδόσεων που δεν το θέσατε. Μπορείτε να μας πείτε αν τα κράτη-μέλη θεωρούν ότι η χρονική στιγμή είναι κατάλληλη για οποιοδήποτε αποθεματικό επιδόσεων. Γιατί είμαστε, γιατί όταν θα φτάσουμε στο ενδιάμεσο σημείο δεν θα μπορούν ε, οι περιφέρειες ή τα κράτη-μέλη να συγκεντρώσουν αυτά τα ποσά. Άρα το, η χρονική στιγμή είναι σημαντική. Το άλλο θέμα που απασχολεί είναι το θέμα της, ε, των πόλεων και των αστικών περιοχών. Μπορείτε να μας πείτε αν τα κράτη-μέλη ανησυχούν για το ποιο θα αποφασίσει για τον ορισμό των πόλεων ή των αστικών περιοχών οι ίδιοι ή θα το αποφασίσουν οι περιφέρειες σημαντικό. Και το τελευταίο αφορά το συνολικό επίπεδο χρηματοδότησης που θα πάει στην πολιτική συνοχής μετά το 2013. Στην αρχική σας δήλωση είπατε ότι τα κράτη-μέλη εκτός ενός ήταν πολύ υπέρ των προτάσεων, αλλά ίσως κάποια κράτη-μέλη να υπάρχει ένα μέρος του προπολογισμού που θα πάει στην ε, Πολιτική συνοχής μετά το 2013. Ποια ε, είναι η επικρατούσα άποψη για λιγότερη ή περισσότερη χρηματοδότηση μετά το 2013. Ευχαριστώ, Φλάσεκ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Υπουργέ, επιτρέψτε μου επίσης να εκφράσω και εγώ τη βαθιά μου ικανοποίηση για τη συνεργασία που είχαμε με την Πολωνική Προεδρία. Διότι μπορούμε να συγκρίνουμε από το πρόσφατο παρελθόν διαδοχικές προεδρίες και νομίζω ότι από την Επιτροπή μας διαπιστώνουμε την προσήλωση στα θέματα που μας ενδιαφέρουν της Πολωνικής Προεδρίας και το αξιολογούμε θετικά. Θα αναφέρω λοιπόν κάποια θετικά στοιχεία και στη συνέχεια θα κάνω μερικές ερωτήσεις. Καλωσορίζω βεβαίως στεναρά ε, τα οικονομικά που προτείνατε ιδιαίτερα για τα νέα κράτη-μέλη. Χαίρομαι που βλέπουμε μια γράμμιση και αύξηση ε, σε σχέση με τη χρήση των πόρων, αλλά ως προς την αποτελεσματικότητα και τις επιδόσεις ακριβώς έχω μια ερώτηση. Γνωρίζουμε ότι σε ορισμένες περιφέρειες έρευσαν χρήματα, ας πούμε, στο Μεσοτζόρνο, στην Νότια Ιταλία, χωρίς να έχει ε, πολύ μεγάλο αποτέλεσμα αυτό η προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που είναι ίδια για όλους είναι σκόπιμη. Ε, ποια θα είναι η συμμετοχή των διαφόρων ταμείων. Μήπως περιορίζουμε την αποτελεσματικότητα, ή υπονομεύουμε ακόμα και τη δυνατότητα ελιγμών που έχουν τα κράτη στην απορρόφηση των κονδυλίων. Προφανώς και δεν θέλουμε να τιμωρήσουμε κανέναν, να αποκλείσουμε κανέναν, αλλά εσείς πώς προτίθεστε να εφαρμόσετε αυτές τις προϋποθέσεις και τους όρους ακριβώς ως προς την πλήρωση και την τήρηση των κριτηρίων. Και μήπως δένουμε τα ίδια μας τα χέρια με τέτοια μέτρα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Υπουργό. Επειδή δεν ε, υποβλήθηκε ερώτηση, στην ε, παρέμβαση του κυρίου Σταυρακάκη. Θα ήθελα να πω ότι το θέμα που θίξατε είναι ένα θέμα το οποίο απασχόλησε την Πολωνική Προεδρία, δηλαδή η ολοκληρωμένη προσέγγιση και το γεγονός ότι θα πρέπει να ασχοληθούμε ιδιαίτερα με την κάθε περιφέρεια. Όπως είπα και πριν, προσδίδουμε μεγάλη σημασία στο κείμενο τη κοινή στρατηγικής πλαισίωσης, γιατί έτσι θα φτάσουμε σε αυτό που δεν είχαμε καταφέρει μέχρι τώρα, δηλαδή τον συντονισμό των διαφόρων πολιτικών. Και το καλύτερο θα ήταν να προσπαθήσουμε να δούμε ποιο είναι το δυναμικό των ευρωπαϊκών περιφερειών. Τώρα, σε σχέση με το θέμα της, ε, την επιφύλαξη ως προς την ε, αποτελεσματικότητα, την απόδοση, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να βρούμε τους ε, πιο ασφαλείς αποτελεσματικούς μηχανισμούς, έτσι ώστε να μπορέσουμε να φτάσουμε στην ύψιστη αποδοτικότητα των προγραμμάτων. Μην ξεχνάμε ότι η τρέχουσα πρόταση της Κομισιόν ενέχει πολλά ενδιαφέροντα στοιχεία, γιατί πρόκειται για ένα εθνικό πλαίσιο και νομίζω ότι θα πρέπει να προωθήσουμε αυτό το αποθεματικό έτσι ώστε να έχει μία κατανομή ανάλογα με τα ορόσημα που ορίζονται και στα οποία ανταποκρινόμαστε είτε ως κράτη-μέλη είτε ως περιφέρειες μέσα στα πλαίσια της απόδοσης μέσα στο πλαίσιο απόδοσης. Έτσι, το νέο αποθεματικό αυτό ασχολείται, επικεντρώνεται περισσότερο στην πολιτική συνοχή, εξ αρχής. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι και στον τρέχοντα υπολογισμό ασχοληθήκαμε με αυτό το θέμα του αποθεματικού. Υπάρχουν πολλαπλές επιπτώσεις, αλλά εξαιτία αυτού του αποθεματικού μπορούμε να είμαστε πλέον αποτελεσματικοί Δηλαδή επικεντρώνουμε την προσοχή μας στα αποτελέσματα και ορισμένα κράτη-μέλη τόνισαν ότι η πρόταση της Κομισιόν ίσως προωθήσει τα εύκολα προγράμματα και θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτό τον κίνδυνο εάν υπάρχει. Σε αντίθεση με τα σχέδια τα οποία είναι και τα καλύτερα και τα πλέον καινοτόμα. Επίσης, αυτό το αποθεματικό ίσως αποθαρρύνει τα θεσμικά όργανα από φιλόδοξους στόχους. Όμως η Πολωνική Προεδρία προσπάθησε να αντλήσει από την θετική της εμπειρία ως προς το αποθεματικό αυτό αποδοτικότητας και με βάση αυτή την γενικότερη όθηση μπορούμε να φτάσουμε σε καλύτερη αποτελεσματικότητα αυτό. Ως προς τον ορισμό της πόλης και του αστικού περιβάλλοντος, την παρούσα στιγμή η συζήτηση για τον ορισμό του άστεως ή της μιας αποκεντρωμένης περιοχής, δηλαδή εκτός άστεως, είναι κάτι που αποφασίστηκε ότι δεν θα τεθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δηλαδή, θα πρέπει να υπάρχουν ορισμοί σε χαμηλότερα επίπεδα. Είναι κάτι παράλληλο, παρόμοιο με το ring fencing, με αυτή την οριοθέτηση που γίνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η ολοκλήρωση. Από όσο γνωρίζουμε, η ολοκλήρωση αυτού του κριτηρίου, η συμπλήρωση αυτού του κριτηρίου δεν είναι κάτι το ευκταίο. Θα πρέπει να γίνει σε κατώτερο επίπεδο. Τώρα ως προς το θέμα του προϋπολογισμού που ετέθη, ως προς τις άτυπες ή μη συναντήσεις, επίσημες συναντήσεις, δεν συζητήσαμε δημοσιονομικά θέματα για το εύρος του προϋπολογισμού. Μιλήσαμε για το πολιετές ε, δημοσιονομικό πλαίσιο. Δεν αναφερθήκαμε καν στο μέγεθος του προϋπολογισμού. Σταθήκαμε στους στόχους, της προτεραιότητες και στο πώς μπορεί να οριστεί καλύτερα αυτή η πολιτική στο μέλλον. Το ερώτημα του κυρίου Βλάσακ ως προς την αυτόματη εφαρμογή ορισμένων παρεμβάσεων σε διάφορα επίπεδα στα πλαίσια δηλαδή του ΕΤΠΑ ή του Ευρωπαϊκού Ταμείου Καινοτόμων Δράσεων, θα πρέπει να καλυφθεί το θέμα μέσω του λεγόμενου ring fencing. Και από τις συζητήσεις φάνηκε ότι αυτό το θέμα αφορά την εταιρική σύμβαση και δεν θα πρέπει να συζητηθεί στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων δεν πρόκειται για ένα ε, αυτόματο επίπεδο το οποίο ορίζεται πανευρωπαϊκά. Ευχαριστώ. Κυρία Πρόεδρε Υπουργέ, θα ήθελα και εγώ να σας ευχαριστήσω για όλες τις πρωτοβολίες ε, που λάνσαρε η Πολωνική Προεδρία. Έγινε πραγματικά συζήτηση επί της ουσίας της πολιτικής συνοχής και τολμώ να πω ότι φτάσαμε σε ένα από τους στόχους που είχαμε θέσει. Η πολιτική συνοχής ε, γίνεται ευρύτατα αποδεκτή στην Ευρωπαϊκή Ένωση με θετικό πνεύμα. Αυτό δεν μπορεί κανείς να το αμφισβητήσει. Στην κατάθεση του νέου νομοθετικού πακέτου της δέσμης αυτής ε, είδαμε ότι ήταν πολύ ευνοϊκή η υποδοχή και συνενετική. Υπάρχουν βέβαια στις οποίες θα πρέπει να επανέλθουμε, αλλά Πρέπει να σας πω, κύριε Υπουργέ, ότι διασκεδάσετε όλες τις αμφιβολίες που είχα πριν ακούσω την τοποθέτησή σας. Έχω όμως και δύο ερωτήσεις. Πρώτον, στο Συμβούλιο, κατά τη διάρκεια της Προεδρίας σας, προσπαθήσατε να βρείτε ποιες πηγές χρηματοδότησης ενδεχομένως να σταματήσουν λόγω των μέτρων ε, που λαμβάνονται για την καταπολέμηση της κρίσης. Να μην θυσιαστεί η ε, πολιτική συνοχή στο βωμό της καταπολέμησης οικονομικής κρίσης. Μπορούμε να βρούμε άλλες πηγές χρηματοδότησης για να μην τα πάρουμε από εκεί. Στη συνέχεια υπάρχει η πολιτική συνοχής και η κοινή γεωργική πολιτική ε, στη δέσμη των μέτρων αυτών. Και θα ήθελα να ρωτήσω, κατά την άποψή σας και κατά την άποψη της Προεδρίας φυσικά γενικότερα, ποια είναι εκείνα τα στοιχεία που μπορούν να μας επιτρέψουν να ενσωματώσουμε την ανάπτυξη της υπαίθρου στην πολιτική συνοχή, να ενοποιήσουμε θέλετε αυτά τα δύο. Έχω ακούσει πολλές απαντήσεις αλλά όχι συγκεκριμένα πράγματα ούτε πιστικά. Εγώ είμαι μέλος ε, και στην Επιτροπή Γεωργίας και εκεί γίνεται μέγας λόγος για την ανάπτυξη της υπαίθρου και τα αντίστοιχα προγράμματα και μάλιστα στο μέλλον θέλουν να τα αποσυνδέσουν από την περιφερειακή ανάπτυξη. Εγώ θέλω την αντίστροφη ακριβώς ε, προσέγγιση. Η ανάπτυξη της υπαίθρου, εξυγχρονισμός της υπαίθρου και των υπαίθριων περιοχών θα πρέπει να συνδέεται περισσότερο με την πολιτική συνοχής. Επίσης πρέπει να σας πω ότι ε, κατά τη διάρκεια του εξαμήνου της Προεδρίας ήταν μια ιδιαίτερη περίοδος αυτή. Τώρα έχει τεθεί σε ισχύ η νέα συνθήκη και βλέπουμε ότι στην εφαρμογή της ε, προκαλούνται διάφορα προβλήματα για σας Υπουργέ και πολλούς από τους συνεργάτες σας και όσους συμμετείχαν σε αυτή την προσπάθεια. Πάντως ε, νομίζω ότι τελικά πήγαν καλά τα πράγματα και σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ λέει Πρόεδρος. Σας ευχαριστώ και εγώ, λέει ο κύριος Τσέλερ, κυρία Υπουργέ, που ξαναβρήκατε το δρόμο προς την Επιτροπή μας. Μάλιστα εσείς ε, το ζητήσατε να έρθετε να μας ενημερώσετε και ευχαριστώ γενικότερα την Βολωνική Προεδρία για την ε, καλή συνεργασία που είχαμε μέχρι σήμερα. Κάτι γενικό που διαπιστώνει κανείς ήταν ότι η Πολωνία ήταν πολύ καλά προετοιμασμένη και πολύ καλά οργανωμένη ε, στην ε, αρχή της Προεδρίας της. Το πρόβλημα μας ε, στη πολιτική συνοχή, στη διαρθρωτική και την περιφερειακή ποιο είναι. Είναι ότι τελειώνει η Πολωνική Προεδρία. Και ο συνάδελφος ο Τσακ είπε πολύ αισιόδοξα ότι η πολιτική συνοχή και η πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι επίμαχες αυτό μπορεί να ισχύει και για την Επιτροπή μας και είναι δικό μας επίτευγμα, αλλά αν κοιτάξω γενικότερα τι γίνεται στο Κοινοβούλιο και στα κράτη-μέλη, στους μη παϊόντες, τα πράγματα αλλάζουν. για αυτά που μας ε, υπέβαλε ως κανονισμό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι αντικείμενο συζήτηση. Στι δύο τελευταίε συνεδριάσει, μάλιστα, συζητήσαμε και εμεί και φαίνεται και σήμερα ότι σε πολλέ από τι προτάσει του κανονισμού έχουμε μάλλον ερωτηματικά παρά απαντήσει που δίδονται. Και εδώ λυπάμαι ακριβώς που μια χώρα όπως η Πολωνία που ε, βλέπει ως κέντρο βάρους και προτεραιότητα την περιφερειακή πολιτική εγκαταλείπει πλέον την Προεδρία. Εγώ δεν θέλω να κατηγορήσω κανέναν, αλλά οι επόμενες δύο προεδρίες νομίζω θα έχουν ε, άλλες προτεραιότητες και όχι απαραίτητο στη διαρθωτική, την περιφερειακή και την πολιτική συνοχής. Και ρωτώ λοιπόν, δώσατε κίνητρα και ενάσματα για τις μελλοντικέ συζητήσεις που σίγουρα θα μας απασχολήσουν ακόμα για πολύ μεγάλο διάστημα και θα μας συνοδεύουν. Δημιουργήστε δομές και οργάνωση στο μέλλον αυτή τη διαδικασία συζήτηση πώς θα την παρακολουθείτε, πώς θα τη συνοδεύετε, γιατί η Πολωνία στο Συμβούλιο έχει κάποιο ειδικό βάρος και ε, σε σχέση με την εσωτερική οργάνωση της πολωνικής κυβέρνησης. Μέχρι τώρα η διασυνοριακή πολιτική και συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών στην Πολωνία ήταν ενταγμένη στο Υπουργείο Εξωτερικών. Και νομίζω ότι μέχρι τώρα αποδείχτηκε γιατί ακούω από την Πολωνία και από τη Γερμανία ότι ενδεχομένω να μην ήταν η σωστή κατάταξη και η περιφερειακή πολιτική στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ακόμα και είναι διασυνοριακή μεταξύ 27 μελών, είναι περιφερειακή πολιτική, δεν είναι εξωτερική πολιτική. Μήπως σκέφτεστε να την απελευθερώσετε εκεί από το Υπουργείο Εξωτερικών για να την αναλάβετε εσείς στο δικό σας Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι τον Ιανουάριο θα έχουμε τον Νικολάη Βάμεν, ο οποίος είναι ο Δανός Υπουργός υπεύθυνο για αυτό το θέμα και για την πολιτική συνοχή. Και από τις συναντήσεις που είχαμε βλέπουμε ότι και η Δανία έχει δεσμευτεί υπέρ αυτής της ε, πολιτικής. είδομεν. Μαρή-Τερέζ Σάντσε-Σμιτ. Ε, σμιτ Ευχαριστώ και σας ευχαριστώ κυρία Υπουργέ για την φιλόδοξη εργασία που προωθήσατε και αναπτύξατε στα πλαίσια της Πολωνικής Προεδρίας για την περιφερειακή πολιτική μιλήσατε για ολοκληρωμένη εδαφική προσέγγιση, ενισχυμένη συνεργασία και νομίζω ότι αν λάβουμε υπόψη τους ε, διάφορους ε, φορείς, εμπλεκόμενους φορείς, μιλάμε για μια πολυεπίπεδη παρέμβαση που να αφορά όλα τα ε, στάδια αυτής της πολιτικής συνοχής. Το θέμα είναι αρκετά συνονιτικό. Υπάρχει μια συμφωνία επί της αρχής. Μέχρι τώρα πόσα μέλη του Συμβουλίου δεσμεύονται επίσημα ε, για αυτή την διακυβέρνηση σε πολλά επίπεδα. Ε, Λάμπερτ Φανίστελ Ρόι, τελευταίος ομιλητής. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ζητώ συγγνώμη που καθυστέρησα και έχασα την ομιλία σας. Έχω όμως μια πολύ μικρή ερώτηση. Για την πολιτική γειτονίας. Γνωρίζω ότι η Πολωνική Προεδρία ενδιαφέρεται πάρα πολύ για τα επιχειρησιακά προγράμματα εκτός των συνόρων και διαπιστώνουμε ότι δεν απέδωσαν ε, όσο θέλαμε κατά τη διάρκεια της περίοδου και θέλησε η Πολωνική Προεδρία να γίνει αυτή η συζήτηση για καλύτερες πρακτικές και μήπως να ξανάρθει στο Ταμείο, το ΦΕΝΤΕΡ της Περιφερειακής Ανάπτυξης, κάποια δράση που είναι στο Ιντερεκ τώρα. Στην τελευταία Ολομέλεια ψήφισε την έκθεση David η ε, Ολομέλεια για την πολιτική γειτονία και το μέλλον της, γενικότερα εκδημοκρατισμός και υποστήριξη των γειτόνων μέσω ΜΚΟ και λοιπά. Σε μία όμως από τις τροπολογίες της δικής μας περιφερειακής πολιτικής της δικής μας Επιτροπής γίνεται λόγος για ενίσχυση του ΦΕΝΤΕΡ στο μέλλον και ενδεχομένω και αυτό το στοιχείο ε, της γειτονίας να βγει από εκεί και να επιστρέψει στην περιφερειακή ανάπτυξη. Το Συμβούλιο πώς το συζητάει, έχετε να μας απαντήσετε τίποτα σχετικά. Υπουργός. ο πρώτος ομιλητής ρώτησε για τις οικονομικές ροές οι οποίες εν δυνάμει θα μπορούσαν να σταματήσουν. Πολλές, έγιναν πολλές ανταλλαγές απόψεων επί του θέματος και αναφέρθηκε και το θέμα των χρηματοπιστωτικών ροών, αλλά δεν θα ήθελα να εξειδικεύσω το θέμα εδώ, αναφερθώ εξειδικευμένα. Ορισμένα κράτη-μέλη αναφέρθηκαν στην μακροαιρεσιμότητα και οι βαλτικές χώρες τάσσονται υπέρ της μακροαιρεσιμότητας ως προς την πολιτική συνοχής. Όμως η μεγάλη πλειοψηφία των κρατών μελών αντιτάχθηκε το να συνδέσουμε τις κυρώσεις με τη μη συμμόρφωση προς τους μακροοικονομικούς δείκτες. Σε σχέση με την πολιτική συνοχής και την μακροοικονομική πολιτική και τους δείκτες, πολλοί από αυτούς που ασχολούνται με αυτό το τομέα είναι πεπισμένοι ότι θα πρέπει να υπάρξει ένας δεσμός μεταξύ της ΚΑΠ και της πολιτικής συνοχής. Βλέπουμε σήμερα ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να θεωρήσουμε τις δύο αυτές πολιτικές ως αυτόνομες οντότητες. Υπάρχει το εταιρικό συμβόλαιο, εταιρικές συμβάσεις που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για να καλύψουν και τις δύο πολιτικές. Όταν μιλάμε με τους ηθήνοντες ε, περί πολιτικής συνοχής, πολλοί λένε ότι η ΚΑΠ ή η αγροτική ανάπτυξη αποτελεί μία μορφή περιφερειακής ανάπτυξης. Άρα θα πρέπει να συνδεθούν οι δύο αυτοί τομείς. Βλέπουμε παράλληλα Είχαμε μία σύντομη συζήτηση και είδαμε ότι υπάρχει διχογνωμία. Αυτοί που ασχολούνται με την ΚΑΠ φαίνεται ότι δεν ασχολούνται τόσο πολύ με την πολιτική συνοχή και δεν βλέπουν αυτό το σύνδεσμο μεταξύ των δύο αυτών πολιτικών. Θα πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι δεν πρόκειται για δύο ξεχωριστές πολιτικές. Και αν ε, μιλούμε για θετικό αντίκτυπο της ε, χρηματοδότησης των περιφερειών ή μίας περιφέρειας συγκεκριμένα θα πρέπει να υπάρχει συμπληρωματικός χαρακτήρας των δύο, κάτι το οποίο δεν ισχύει μέχρι σήμερα. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τα ε, θετικά σας λόγια για το έργο της Πολωνικής Προεδρίας. Θα ήθελα επίσης να πω προς την Πρόεδρο ότι θα εκπλαγείτε θετικά και με τα αποτελέσματα το έργο της Δανέζικης Προεδρίας. Γιατί έχουμε συνεργαστεί εκ του σύνεγγης με τη Δανία μέσα στα πλαίσια των τριών προεδριών και είχαμε συζητήσεις εξ αρχής και με την ε, μελλοντική προεδρία, την Προεδρία της Δανίας. Δεν θα πρέπει να προδικάσουμε λοιπόν την κατάσταση σήμερα, διότι πιστεύω ότι τα αποτελέσματα θα είναι ιδιαίτερα θετικά. Αυτή είναι η γνώμη της Πολωνικής Προεδρίας. Με την ευκαιρία αυτή θα ήθελα να αναφέρω ότι με βάση τα σημερινά δεδομένα βλέπουμε ότι υπάρχουν διαφορετικές απόψεις από τις μεμονωμένες κυβερνήσεις. Όταν συζητούμε στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων, είδαμε ότι συμμετείχαν και υπουργοί από άλλα υπουργεία και είδαμε ότι υπήρχε ομοφωνία Είδαμε λοιπόν ότι άλλοι υπουργοί από το ίδιο κράτος μέλος μας ε, προέβαλαν μια διαφορετική ιστορία. Η Δανία νομίζω δεν αντιμετωπίζει αυτό το θέμα. Πιστεύω λοιπόν ότι οι μελλοντικές εξελίξεις θα είναι θετικές. Θα συνεργαστούμε με την Προεδρία, τη μελλοντική Προεδρία της Δανίας όπως έγινε και μέχρι τώρα. Η κυρία Σάντσες Σμιτ υπέβαλε ένα ερώτημα σε σχέση με, την, με το περιφερειακό επίπεδο και το γεγονός της αποκέντρωσης που χρειάζεται. Όλα τα κράτη-μέλη συνειδητοποιούν τη σημασία του περιφερειακού και τοπικού επίπεδου ιδιαίτερα ως προς τα άστεα. Όμως δεν έγινε μία συζήτηση μέχρι τούδε για την συμπερίληψη των περιφερειακών κυβερνήσεων στο, στο, στις εταιρικές αυτές συμβάσεις. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρξει συνεργασία σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, αλλά δεν έχει δοθεί οριστικός χαρακτελικός χαρακτήρας Το Βέλγιο ήταν η μόνη χώρα που μίλησε για τις περιφέρειες που θα πρέπει να συμπεριληφθούν σε αυτό το θέμα και προς τον κύριο Βανίστελ Ρόι. Θα ήθελα να πω ότι πράγματι, απαντώντας στην ερώτηση της κυρίας Μάνερ, που μου μίλησε για την εδαφική ε, συνεργασία, μίλησα εκτενώς, απάντησα εκτενώς επί του θέματος. Ε, ίσως τώρα μπορώ να σας πω και κάτι άλλο. Μας απασχολεί και η πολιτική γειτονίας και η κοινή αυτή εργασία με τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις γείτονες χώρες. η εμπειρία μας, από, την, από τις εμπειρίες μας, μπορούμε να πούμε ότι τα δεδομένα είναι αρκετά αρνητικά. Εάν τα προγράμματα αυτά ακολουθήσουν ως έχουν ως προς την πολιτική γειτονία, ίσως αντιμετωπίσουμε προβλήματα για την δαπάνη των κονδυλίων. Η Φινλανδία άρχισε μία εκτεταμένη ε, εργασία επί του θέματος και θα δούμε ποια θα είναι η εξέλιξη. Ο Νίκολας Μάρτιν από την Επιτροπή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω καταρχήν με την ευκαιρία αυτή να ευχαριστώ την κυρία Υπουργό για την προσωπική της αφοσίωση στην πολιτική συνοχής η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη εκτιμήσει ιδιαίτερα τα επιτεύγματα που έγιναν δυνατόν να έχουμε λόγω της δικής της ε, αφοσίωσης και των συνεργατών της. Σε χρόνο ρεκόρ έγιναν οι δύο τροποποίησεις των δύο κανονισμών που ήταν απαραίτητες και ακριβώς χάρη στην ε, στοχευμένη προσπάθεια της Προεδρίας και την αφοσίωση της Επιτροπής σας και της Προέδρου επιτεύχθηκαν όλα αυτά. Και αυτό αποδεικνύει το τι μπορεί να γίνει όταν πράγματι υπάρχει πολιτική ανάγκη να γίνει κάτι. Επίσης εκτιμάμε τον τρόπο με τον οποίο ε, μπόρεσε να αναπτυχθεί η συζήτηση για την εδαφική διάσταση σε διάφορους χώρους, όπως είπε και ο υπουργό. Θεωρώ ότι αυτό αποτελεί σε καλή βάση για τη συζήτηση της πολιτικής συνοχής και το θέμα της σχέσης ανάμεσα στην εδαφική διάσταση της πολιτικής και το στόχο του 2020. Θεωρώ ότι η πρόοδος που έχει επιτευχθεί στο πλαίσιο του νομοθετικού πακέτου είναι εντυπωσιακή δεδομένου του περιορισμένου χρόνου. Και έχω προσωπικά υποφέρει, αλλά πρόθυμα υποφέρει λόγω της εντατικής εργασίας, δεδομένου ότι πραγματικά χρειάζεται η, η ταχεία πρόοδος. Υπάρχουν σημαντικά σημεία όπου έχει γίνει πραγματικά ενδελεχής δουλειά, η οποία αποτελεί εξαιρετική βάση για την Δανέζικη Προεδρία η οποία θα μπορέσει να προχωρήσει. Και βεβαίω και στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων τη Παρασκευή έγινε συζήτηση. Εκτιμήσαμε το γεγονό ότι έγινε Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων ειδικά για την πολιτική συνοχή. Αυτό επέτρεψε να γίνει μια σωστή συζήτηση και να έχουμε χειροπιαστά αποτελέσματα. Δύο λόγια τώρα για τα τρία βασικά ζητήματα που αποτελούν θεμελιώδη ζητήματα ε, στη συζήτηση για το νομοθετικό πακέτο, για το πακέτο των κανονισμών και για την Επιτροπή. Στο κοινό στρατηγικό πλαίσιο. Εμείς από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής θεωρούμε ότι πλέον η έμφαση πρέπει να δοθεί στην ανάπτυξη του περιεχομένου του κοινού πλαισίου, ώστε να ξεκαθαρίσουμε αν υπάρχει κοινή άποψη για το πώς θα επιτευχθεί η προστιθέμενη αξία του εγγράφου. Όπως γνωρίζετε, ε, δουλεύουμε σε ένα, πάνω σε ένα σχέδιο του εγγράφου, το οποίο θέλουμε να μπορέσουμε να παρουσιάσουμε για να δοθεί ευκαιρία να ακούσουμε απόψεις και του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου. Να διαπιστώσουμε αν υπάρχει κοινή προσέγγιση για το πώς θα επιτευχθεί και το στρατηγικό στοιχείο, αλλά τελικά θα έχουμε και ένα χρήσιμο έγγραφο που θα επιτύχει το στόχο του ή θα αποτελεί σημείο αναφορά για τις, ε, τα κράτη-μέλη που θα προετοιμάζουν τα, τις ε, συμβάσεις εταιρική σχέση κλπ. Στο πλαίσιο αυτό θεωρούμε ότι θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε για την διαδικασία έγκρισης. Το δεύτερο ζήτημα ε, προτάσεων που είναι συγκεκριμένες για κάθε χώρα. Αυτές, αυτές έχουν σχέση με το μηχανισμό σύνδεσης του, της πολιτικής συνοχής με την πολιτική του 2020. Αυτό παραλήφθηκε και στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων. Και το ζήτημα είναι πώς θα θεσπιστεί ένας σωστός μηχανισμός για να επιτευχθεί αυτό. Η άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι ότι οι συστάσεις θα αφορούν την κάθε χώρα συγκεκριμένα, θα πρέπει να είναι κομμάτι της όλης διαδικασίας γιατί εντάσσονται στον υφιστάμενο μηχανισμό της ε, υλοποίησης στρατηγικής Ευρώπης 2020. Υπάρχει λοιπόν η πρέπει να υπάρχει διαβεβαίωση ότι τα εθνικά προγράμματα μεταρρύθμισης των κρατών μελών θα συνεισφέρουν στην επίτευξη αυτών των προτεραιοτήτων. Αν δεχτούμε ότι η πολιτική συνοχή θα είναι σημαντική στο να συνεισφέρει ε, οικονομικά στην επίτευξη των προτεραιοτήτων και των στόχων της Ευρώπης 2020, θα πρέπει να δεχτούμε και ότι η συστάσεις για κάθε χώρα θα, παίξουν, θα παίξουν το ρόλο του. Από πλευρά Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα είναι αδιανόητο η διαδικασία και τη προετοιμασία των προγραμμάτων και των ε, συμβάσεων σχέση σχέση κρατών μελών θα γίνουν χωρί να ληφθούν υπόψη οι συστάσει ε, που είναι ειδικέ για κάθε χώρα και ούτε μπορεί να τι ε, αγνοήσει αυτέ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γι' αυτό πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι οι μηχανισμοί που θα συσταθούν θα κάνουν τη σύνδεση αυτή. Και πράγματι αυτό είναι ένας από τους στόχους του, που θα, πρέπει, θα μπορεί να παίξει το κοινό στρατηγικό πλαίσιο. Να δείξει πώς μπορεί να αναπτυχθεί αυτή η σχέση. Στο θέμα τώρα της θεματικής συγκέντρωσης και πάλι υπάρχει μια ευρεία συνένωση ότι πραγματικά υπάρχει αυτή η ανάγκη. Αλλά έχουμε και ενδείξεις ότι υπάρχει ανάγκη για ευελιξία. Δεν είναι όμως απόλυτα σαφές το πώς θα επιτεθεί αυτή η ευελιξία. Η στάση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι ότι υπάρχει ακόμα περιθώριο να διερευνηθούν ε, να διερευνηθεί η εφαρμογή στην πράξη του μηχανισμού των διαφόρων ταμείων και ότι δεν έχουμε ακόμα αντιληφθεί πλήρως τις δυνατότητες ευελιξίας που προσφέρουν αυτοί οι μηχανισμοί και ότι επίσης μπορούμε με ένα χρήσιμο τρόπο και πρακτικό να δούμε πού υπάρχουν συγκεκριμένες ανάγκες για ευελιξία ώστε να επιτευχθούν δαφική, συγκεκριμένη στόχη. Δηλαδή στις περιπτώσεις όπου αν λείπει αυτή η ευελιξία θα προκύψουν κάποιες ανομαλίες. Έτσι λοιπόν ήταν χρήσιμο που έγινε αυτή η συζήτηση, η οποία όπως και οι συζητήσεις της ομάδας εργασίας του Συμβουλίου θα αποτελέσει τη βάση για περαιτέρω πρόοδο στη διάρκεια της Προεδρίας Δανίας. Ένα άλλο, μια σειρά από άλλα θέματα ετέθησαν στη διάρκεια της συζήτησης κυρία Πρόεδρε και είμαι βέβαιος ότι θα μπορέσουμε αργότερα να τα θέσουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Νίκολας. Καταλαβαίνω από αυτά που λες ότι υπάρχουν διστάμενες απόψεις για κάποια θέματα σήμερα. Και αυτό για το Κοινοβούλιο είναι σημαντική πληροφορία. Αυτό το κομμάτι της παρουσίασής σου μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε και ως εισαγωγή στο επόμενο θέμα. Εν πάση περιπτώσει, στη φάση αυτή θέλω να πω εκ μέρους όλων μας της Επιτροπής αυτών και ε, αυτών που δεν έχουν έρθει γιατί έχουν αρχίσει τις γιορτέ, να γιορτάζουν τα Χριστούγεννα στα σπίτια τους, ότι εκτιμήσαμε ιδιαίτερα τη συνεργασία και ότι πραγματικά ε, εκτιμήσαμε ιδιαίτερα την τον εντατικό ρυθμό της δουλειάς σας, γιατί μεταξύ της 6 Οκτωβρίου που θέσπισε το ρυθμιστικό πλαίσιο η Κομισιόν και της 16 Δεκεμβρίου που έγινε το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων για την ανακεφαλαίωση είναι δύο μήνες και λίγες μέρες και πραγματικά έγιναν πολλά στο διάστημα αυτό και ελπίζουμε ότι με την ίδια ταχύτητα θα συνεχίσουμε και τους επόμενους μήνες. Θέλω λοιπόν να σας ευχαριστήσω ιδιαίτερα κυρία Υπουργέ για την ε, συνεισφορά σας, για την συμμετοχή σας και θα πρέπει πιστεύω να ε, περιμένουμε να συνεχίσετε να εμπλέκεστε και στο μέλλον, μέλλον λόγω της ε, εμπειρίας που έχετε αποκτήσει να συνεργαστείτε με τις μελλοντικές προεδρίες. Θέλω λοιπόν να σας δώσω για ένα λεπτό ακόμα το λόγο να μας αποχαιρετήσετε. Uh, thank you very Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους για τη συνεργασία ελπίζω μέσα στα πλαίσια της ε, τριμερούς ε, συνάντησης των προεδριών, των τριών προεδριών, να έχουμε πολύ καλή συνεργασία και με την Προεδρία της Δανίας. Σας εύχομαι καλά Χριστούγεννα και όλα να πάνε καλά για όλους. Σας ευχαριστώ πολύ. One, one minute to say goodbye to Μια αποχαιρετήσω την Υπουργό. Λοιπόν, σε δύο λεπτά αρχίζει το επόμενο θέμα. Θα ήθελα να αξιοποιήσω αυτό το δίλεπτο για να σας ε, κάνω τις ανακοινώσεις Προέδρου. Το σημείο 10 στην ημερησία διάταξη είναι η τροποποίηση του κανονισμού ε, για τα μέσα επιμερισμού του κινδύνου. Σήμερα δεν μπορεί να γίνει συζήτηση διότι η δυναμική ε, της διαδικασίας δεν μας επιτρέπει να έχουμε ουσιαστική συνεδρίαση και ανταλλαγή απόψεων σήμερα. Γι' αυτό θα σας πρότεινα να γίνει την επόμενη φορά, στην επόμενη συνεδρίαση. Ε, στο μεταξύ αναβλήθηκε η συζήτηση και στο Συμβούλιο και δεν ε, συζητήθηκε στις 15 Δεκεμβρίου, αλλά θα γίνει αύριο. Επίσης, Σήμερα το πρωί είχε προγραμματιστεί να συναντηθούν όλοι οι θεσμοί και τα θεσμικά όργανα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, δικοί μας ηγητές και όδης, Δανική Προεδρία, Πολωνική Προεδρία. Δεν έλαβε χώρα ε, αυτή η συνεδρίαση γιατί οι περισσότεροι έλειπαν. Αυτή η τεχνική λοιπόν συνεδρίαση για να καταλάβουμε καλύτερα τι προτείνεται θα γίνει στις 11 του μηνός Ιανουαρίου και η δική μας συνεδρίαση είναι στις 25 και 26 ε, Ιανουαρίου, οπότε εκεί μπορούμε να ανταλλάξουμε απόψεις για τα όσα θα έχουν διαμειφθεί και τη νέα πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Λοιπόν, αυτές ήταν οι ανακοινώσει μου. Προχωρούμε λοιπόν στο επόμενο θέμα της μέρης της διάταξης που είναι δεύτερη συζήτηση στην Επιτροπή μας για αυτό που ονομάζουμε γενικό κανονισμό. Η σημερινή συζήτηση βασίζεται και πάλι στο έγγραφο εργασίας που λάβατε για τη συνεδρίαση της 14ης ε, Νοεμβρίου και εγγράφεται στα πλαίσια των όσων είχαμε συμφωνήσει με τους δύο εισηγητές, αλλά να δώσω το λόγο και στους δύο, δεν ξέρω με ποια σειρά, πρώτος ο Λάμπερτ και μετά η Κωνσταντσε η Κωνσταντζή σου λέει να πάρεις εσύ πρώτο το λόγο, ορίστε. Αν θες να κάνεις εσύ τα εισαγωγικά σου σχόλια, παρατηρήσεις, παρακαλώ. Το κάνουμε ξανά και ξανά, αλλά πάντοτε μπερδεύουμε για το πιανού σειρά είναι. Είναι η δική μου σειρά. Τώρα, επί της διαδικασίας. Είναι απολύτως σαφές ότι ήδη την προηγούμενη φορά έγινε μια πρώτη εισήγηση και 11 θέματα, 11 σημεία, τα οποία αποτελούν τα βασικά σημεία που πρέπει καταρχήν να συζητηθούν πριν ε, γίνει η ακρόαση και έχουμε να αντιμετωπίσουμε τροπολογίες. Αυτή τη φορά ίσως μας δοθεί η δυνατότητα να ακούσουμε περισσότερα σχόλια από τους συναδέλφους. Την προηγούμενη φορά ήμασταν λίγο περιορισμένοι από το χρόνο είχαμε και τους εισηγητές των τριών, τεσσάρων ε, κανονισμών που εμπλέκονται εδώ. Χρειάστηκε λοιπόν να ακούσουμε, θα θέλαμε λοιπόν να ακούσουμε περαιτέρω σχόλια. Τι έγινε η αλλαγή. Την προηγούμενη φορά ε, ασχοληθήκαμε με τέσσερα σημεία για να τα διευκρινίσουμε μετά θα άλλα 3-4 και μετά τα τελευταία 3-4 και θα έχουμε φτάσει πλέον στη στιγμή της ακρόασης και θα πάμε στη φάση ε, της τροποποίησης. Αυτή τη φορά ήταν το 1 και είμαστε πολύ σαφείς εδώ στην, στην Επιτροπή μας για το κοινό στρατηγικό πλαίσιο. Η άποψή μας είναι ότι πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του, της νομοθετικής διαδικασίας, της συνομοθετικής διαδικασίας του Κοινοβουλίου. Ίσως να το κάναμε χωριστό κανονισμό ή παράρτημα του κανονισμού αυτού. Αυτό μπορεί να συζητηθεί περαιτέρω. Όμως, Αυτές είναι, θέμα, το θέμα που μας απασχολεί και είναι θετικό ότι η νομική υπηρεσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατέληξε ότι η, θα πρέπει να τηρείται η συνήθις νομοθετική διαδικασία και χαιρόμαστε που η πρόεδρος της Επιτροπής έχει ήδη προωθήσει μια επιστολή με το αίτημα αυτό προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή την οποία ζητάει αυτή την προσέγγιση. Υπάρχουν τρία ε, ερωτήματα εδώ, λεπτομερές, ε, κάποιες λεπτομέρειες πώς να δούμε το θέμα. Ε, βλέπετε ποια είναι τα σημεία. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που το Συμβούλιο, μόλις ακούσαμε ότι έστειλε τις ίδιες επιθυμίες για την αναβάθμιση, θα μπορούσα να πω, του κοινού στρατηγικού πλαισίου από κατεξουσιοδότηση πράξης σε κανονική ε, νομοθετική διαδικασία. Αυτό είναι το πρώτο. Ελπίζω ότι θα το κερδίσουμε. Μόλι άκουσα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι είναι διατεθειμένη να παρουσιάσουν ένα έγγραφο, αλλά δεν είναι σωστή αυτή η σειρά. Υπάρχει τέτοια ξεκάθαρη άποψη από πλευρά Κοινοβουλίου Ίσως θα πρέπει οι νομικοί να έρθουν σε επαφή μεταξύ τους, αλλά για τους πολιτικούς το, το αποτέλεσμα είναι ξεκάθαρο. Είναι κάτι που πρέπει να γίνει. Δεύτερον, είναι τα... Ε, οι συμβάσεις εταιρική σχέσης. Εδώ υπάρχει κάτι που ενδεχομένως μπορούμε να το δεχτούμε ως ε, την άποψη των εισηγητών. Την προηγούμενη φορά μας εξήγησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι θα πρέπει ιδιαιτέρως να αντιμετωπιστεί αυτό ως ένα έγγραφο εκ των κάτω προς τα άνω και όχι απλώς το αντικείμενο διαπραγματεύσεων μεταξύ κρατών μελών κυβερνήσεων δηλαδή και Ευρωπαϊκής Επιτροπής, είναι ένα έγγραφο που στηρίζεται ε, στην προσέγγιση όπου εμπλέκονται όλα τα επίπεδα, όλοι οι εταίροι. Και μπορούμε να δεχτούμε κάποιες από τις προηγούμενες ιδέες μας, ώστε να υπάρξει ξεκάθαρος ορισμός πριν καν ξεκινήσουμε για το ποιοι είναι οι εταίροι και ποια είναι η... θα πρέπει να είναι αυτή η συμβατική σχέση. Αυτό είναι το δεύτερο σημείο, υπάρχουν τα λεπτομερή... λεπτομέρειες εκεί. Επίσης, ακούσατε πριν από λίγο ότι από το σημείο 3 γίνεται κάτι. Πρέπει όμως να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι για τις θεματικές προτεραιότητες και για την ευελιξία που προσφέρεται. Επειδή, όπως γνωρίζετε, η πολιτική συνοχής ε, έχει περισσότερα στοιχεία ε, στην προσέγγιση της και στη δομή της από ότι η Ευρώπη του 2020. Υπάρχει αυτή η επιπλέον εδαφική διάσταση που ε, λαμβάνεται υπόψη Ίσως και εδώ προσφέρω κάποια ευελιξία στην Κόνσταντς. Ε, έχει πολύ συγκεκριμένες ιδέες για να προωθήσει την ευελιξία. Δεν ξέρω αν τώρα η κατάλληλη στιγμή, Κωνσταντ. Ναι, ευχαριστώ πολύ, Λάμπερτ, για την πρώτη εισαγωγή αυτή. Αγαπητοί συνάδελφοι, διαπιστώνεται ότι η συζήτηση που έχουμε με όλους εκπροσώπους και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την Προεδρία, αλλά και άλλους εκπροσώπους συμφερόντων των περιφερειών, έχει προχωρήσει πάρα πολύ η συζήτηση που έχουμε οι δύο εισήγητες και έχουμε πει σε πιο συγκεκριμένα πράγματα πλέον στο έγγραφο εργασίας. Το πρόβλημα ποιο είναι. Όσο βαθαίνει κανείς στη συζήτηση, διαπιστώνουμε ότι θεματικές προτεραιότητες, η ευελιξία, οι και οι συμβάσει εταιρικέ σχέσεις είναι πάρα πολύ στενά συνδεδεμένα μεταξύ τους στους θέματα. Και όταν τραβήξεις κάπου μια κλωστή, ε, ξυλώνεται κάπου αλλού μια ολόκληρη ε, κατάσταση. Θα πρέπει να το μελετήσουμε σε μεγάλες λεπτομέρειες. Μέχρι τα τέλη του έτους, νομίζω, πρέπει να φέρουμε στη συζήτηση κάποια συγκεκριμένη πρόταση. Κάποια στιγμή όλα αυτά θα πρέπει να αποκρισταλωθούν και να πούμε ότι ως Επιτροπή καταρχάς και στη συνέχεια ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέλουμε να ακολουθήσουμε μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Το διαβλέπετε ήδη στις ερωτήσεις Στη συμβάση εταιρική σχέση θα θέλαμε πολύ εντονότερη συμμετοχή των περιφερειών. Το πώς οργανώνεται αυτό από νομικής πλευράς, εντάξει κάθε χώρα λειτουργεί διαφορετικά, η συνταγματική δομή και συγκρότηση κάθε χώρας διαφέρει. Ούτε είναι η δική μας δουλειά, δεν χρειάζεται εμείς να το εξακριβώσουμε αυτό ή να το διευκρινίσουμε. Αυτό είναι θέμα των νομικών υπηρεσιών. Η πολιτική βούληση είναι όμως να επιτευχθεί πολύ μεγαλύτερη συμμετοχή των περιφερειών για να αντιμετωπίζονται οι ειδικέ ε, ανάγκες της κάθε περιφέρειας και με τρόπο δεσμευτικό στις συμβάσεις για την εταιρική σχέση. Προς τα εκεί πιστεύω θα πρέπει να στραφούμε. Αν το πράξουμε έτσι και αν βάλουμε και ένα στίγμα, θα μπορούσε κανείς να πει ναι στις θεματικές ενότητες και στη συγκέντρωση, αλλά με πολύ πιο έντονη συμμετοχή των περιφερειών και να επιλέγουν εκείνες. Βεβαίω πάντα υπό την επικεφαλίδα στρατηγική 2020 αλλά και πολιτική συνοχή. Τι ε, θεωρούν ιδιαίτερα σημαντικό οι περιφέρειες να έχουν την ευκαιρία εκείνες να ορίζουν καλύτερα και να εκφράζουν καλύτερα τις ανάγκες τους. Στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις θεματικές προτεραιότητες γίνεται λόγος για κάτι που πιστεύω πρέπει να μας απασχολήσει και μας. Νομίζω ότι λείπουν ένα-δύο πράγματα και τις τελευταίες εβδομάδες και μήνες ακούμε πολύ συχνά τη δημογραφική εξέλιξη ως όρο. Μάλιστα ολόκληρη έκθεση είχαμε πρόσφατα και στο Κοινοβούλιο σχετικά. Θα μπορούσα να φανταστώ να πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι εντάξει όλα αυτά τα έχετε συμπεριλάβει στις προτεραιότητες που αναφέρονται, αλλά νομίζω ότι ως βασική και οριζόντια απέτηση θα πρέπει να αναφέρεται αυτό παντού. Το έχουμε και στην τωρινή προγραμματική περίοδο, όταν ε, την προετοιμάζαμε, το συζητήσαμε εντατικά. Υπάρχει έτσι και γενικά και αόριστα και συγκεκριμένα σε διάφορα προγράμματα, κανονισμούς κτλ. Αλλά δεν νομίζω ότι μεταφράζεται αυτό στην πράξη σε συγκεκριμένα έργα, προγράμματα, ανάπτυξη της περιφέρειας. Γι' αυτό πιστεύω ότι είμαστε υποχρεωμένοι και θα πρέπει να αναλάβουμε και την ευθύνη αυτή να στείλουμε ένα μήνυμα πιο σαφές. Ότι η μελλοντική ανάπτυξη δεν θα πρέπει να είναι μόνο αϊφόρους και να εξοικονομεί πόρους από πλευράς περιβάλλοντος και κλίματος, αλλά θα πρέπει να ασχολούμαστε ε, και με τρόπο πιο αηφόρο και πιο προσεκτικό με τους ανθρώπους. Να κοιτούμε προς τα πού ε, αναπτύσσεται ο πληθυσμός στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι θα χρειαστεί στο μέλλον ως υποδομές. Ενδεχομένως τι να μην χρειάζεται πια. Παράδειγμα. Στον κανονισμό γίνεται μια πολύ ομοία αναφορά ότι δεν επιτρέπονται πλέον προγράμματα υποδομών στις καλύτερα ανεπτυγμένες περιφέρειες. Και αυτό χωράει συζήτηση. Δεν νομίζω ότι είναι χρήσιμο ε, ρητά σε έναν κανονισμό να απαγορεύεται με τέτοιο ομό τρόπο οποιαδήποτε υποδομή χωρίς να έχουν ούτε κατά διάνοια ε, τη δυνατότητα οι περιφέρειες να εξηγήσουν για ποιο λόγο χρειάζονται ενδεχομένω ορισμένες ε, υποδομές. Το θεωρώ αυτό πολύ δύσκολο να περάσει. Ιδιαίτερα όταν ακούμε για υποδομές και για μέτρα, οι περισσότεροι μπορούν να σκέφτονται τα έργα οδοποιίας, αλλά οι υποδομές δεν είναι μόνο οι δρόμοι, είναι πολύ περισσότερα. Ιδιαίτερα όταν μιλούμε για νέες προσεγγίσεις στην ενεργειακή πολιτική, ακριβώς και οι ανανεώσιμες είναι προτεραιότητα και η ενισχυσή τους, τότε θα μπορούσαμε να ξέρουμε ότι αυτό σημαίνει και αποκεντρωμένη διανομή της ενέργειας. Χρειάζεται δηλαδή να ε, κάνουμε επενδύσεις σε δίκτυα. Και δεν καταλαβαίνω γιατί θα πρέπει ρητά να απαγορεύεται οποιαδήποτε επένδυση σε υποδομές, να το ξανασυστήσουμε αυτό οπωσδήποτε. Είναι και αντιπαραγωγικό κατά τα άλλα. Για την ατζέντα της Ένωση το 2020. Το τέταρτο σημείο της ευελιξίας και των ποσοστώσεων, το είπα και την περασμένη φορά, ειλικρινά δεν έχω προχωρήσει πολύ. Δεν έχω έτσι επισκόπηση πόσες φέτες από ποια ταμεία χρησιμοποιούνται για ποιο σκοπό. Γιατί όσο πιο προσεκτικά και από κοντά τα κοιτάει κανείς, τόσο περισσότερο συγκεχημένη είναι η εικόνα νομίζω θα πρέπει να το συζητήσουμε από κοινού. Δεν είναι μόνο στο γενικό κανονισμό, είναι σε όλους τους κανονισμούς για όλα τα ταμεία. Και θα πρέπει να το συζητήσουμε πιο εντατικά, εάν και κατά πόσο είναι απαραίτητο από την αρχή να έχουμε προσημείωση, earmarking ή ποσοστώσεις. Από πλευράς δημοσιονομικής θα επιτρέπει ε, για την πολιτική συνοχή της περιφέρειας μόνο ένα 10% του ποσού. Πρέπει οπωσδήποτε να το κοιτάξουμε αυτό πιο εντατικά. Θα μπορούσα να σας κάνω και προτάσεις εδώ αν θέλετε. Οι μεν θα χαρούν, οι δε θα εκνευριστούν φρικτά, οπότε επειδή είναι και Χριστούγεννα τώρα, μην κάνουμε τέτοιες συζητήσεις, να πάμε να ξεκουραστούμε. Ε, θα το συζητήσουμε και με τον Λάμπερτ Βανίσε Ρόι και αρχές του επομένου έτους που θα έχουμε μαζέψει δυνάμεις θα μπορέσουμε από κοινού να ξανασυζητήσουμε τις πιο αισιόδοξε ε, εναλλακτικέ και μεταβλητέ για την, για την περιφερειακή πολιτική και την πολιτική συνοχή. Βασιζόμαστε στη σοφία σας και πιστεύουμε τα Χριστούγεννα θα είναι καλό σύμβουλο. Θα, δώσουμε, θα δώσω τώρα το λόγο στους σκιώδεις και στη συνέχεια στα μέλη της Επιτροπής. Ποιος θα ήθελε το λόγο σας, παρακαλώ να σηκώσει το χέρι. Δεν ξέρω κατά πόσο ο κύριος Κούντμαν θα ήθελε το λόγο. Ο σκιώδης έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ για τη δυνατότητα αυτή που μου δίνετε. Έχω σχόλια από τη δική μου πλευρά. Νομίζω ότι δεν είναι εύκολο να έχω άμεσες απαντήσεις. Ως προς το πρώτο θέμα που έφεξε ο κύριος Βανίστελ Ρόι, τι θα γίνει με το κοινωνικό ταμείο, θα παραμείνει στα πλαίσια της πολιτικής συνοχής ή όχι. Αυτό θα πρέπει να το επεξηγήσουμε σαφώς διότι έχουν αναλυφθεί περισσότερες πρωτοβουλίες να περάσει το εκταλού. Πιστεύω όμως ότι θα πρέπει να γίνει να μην... Δεν ξέρω κατά πόσο πρέπει να γίνει αυτή η αλλαγή, αλλά θα πρέπει να δούμε τι επιπτώσεις έχει καταρχήν. Το δεύτερο θέμα αφορά την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση. Φαίνεται, διακυβέρνηση φαίνεται και στις μικρότερες χώρες η δημοκρατία είναι μια πάγια δομή η οποία αφορά όλα τα επίπεδα. Στα πλαίσια της πολιτικής συνοχής, δεν ξέρω σε ποιο επίπεδο βρίσκονται στο ΝΑΤΣ 1 ή στο ΝΑΤΣ 2. Υπάρχει μεγάλη ε, διαφορά στη δική μου χώρα μεταξύ ΝΑΤΣ 1 και ΝΑΤΣ 2. Θα πρέπει στο επόμενο πλαίσιο να ε, έχουμε το ίδιο σύστημα, δηλαδή να έχουμε τα τετραγωνικά χιλιόμετρα όπως ορίζονται μέχρι τώρα. Μέσα στα πλαίσια του ΕΤΠΑ, οι περιφερειακές δομές που υπάρχουν θέλουν να διαδραματίσουν διαφορετικό ρόλο. Εδώ μιλώ για τα ε, δημοτικά συμβούλια. Δηλαδή, ε, όπως ξέρετε, η Λετωνία είναι μία περιφέρεια. Θα πρέπει να παραμείνουμε με αυτή τη συγκεκριμένη δομή, αυτή τη διάρθρωση. Ως προς το θέμα το υπαριθμών 3, σε σχέση με τις ε, θεματικές ε, εναλλακτικές λύσεις, σε σχέση με την πολιτική 2020, έχουμε υποβάλει αρκετές ε, προτάσεις προς την Κομισιόν. Δεν πρόκειται για ένα μεγάλο, μια μεγάλη ποσοστή αναλογία των προτάσεών μας μέσα στα πλαίσια του 2020, αλλά μας ενδιαφέρουν οι μακροχρόνιες πολιτικές της πολιτικής συνοχής, διότι ίσως μετά το 2020 να έχουμε, τι να έχουμε, το 3030, τι θέλετε. Αυτό που θα πρέπει να κάνουμε είναι να ε, συμφωνήσουμε Δηλαδή αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να δούμε τη συνοχή έτσι ώστε αυτοί που βρίσκονται σε χαμηλότερο επίπεδο να ενταχθούν στο πλαίσιο συνοχής και μετά να περάσουμε σε ανώτερο ε, επίπεδο, δηλαδή να κινηθούμε από κοινού. Σε σχέση με την ευελιξία και τις ποσοστώσεις, αυτό δεν είναι τόσο σαφές ε, για μένα, διότι αν μιλάμε για ευελιξία, θα πρέπει να δούμε τι γίνεται Ω ως προς την προϋπάρχουσα κατάσταση. Δηλαδή θέλουμε να είμαστε ευέλικτοι μέσα στα πλαίσια ενός ταμείου. Δηλαδή, αν κανείς δεν τηρεί τις υποχρεώσεις του σε ένα ταμείο, δεν μπορεί να περάσει ένα άλλο. Και είναι πολύ δυσκολότερο για τους δικαιούχους να αλλάξουν κατάσταση. Ίσως έχουν ενταχθεί στο έτπα ή σε μια διαφορετική πολιτική συνοχή. Σε πάση περιπτώσει έχουν σταματήσει. Θα θέλαν λοιπόν να αλλάξουν, να περάσουν σε ένα άλλο πλαίσιο. Μιλάμε για τέτοιου είδους ευελιξία. Ε, κάπου θα πρέπει να ενταχθεί αυτό. Θα πρέπει να τονιστεί ότι όταν εργάζεται κανείς ε, σε ένα ταμείο, έχει ενταχθεί σε ένα ταμείο, δεν θα πρέπει επειδή τα πράγματα ε, δεν πάνε καλά να ζητήσει να μετατεθεί σε ένα άλλο ταμείο. Βεβαίως, έχουμε, έχουμε μιλήσει ως προς τις ποσοστώσεις, έχουμε μιλήσει για αλλαγές σε σχέση με τις οροφές, αλλά δεν ξέρω ποια είναι η διαφορά. Εάν υπάρχουν υποχρεωτικές ποσοστώσεις, Μπορεί να υπάρχουν δυνατότητες μέσα στα πλαίσια του 2,5% να είμαι επιτυχής. Αν δεν είμαι, τι είναι, ποιες είναι οι ποσοστώσεις που εντάσσονται σε αυτό το ανώτατο όριο. Εξηγήστε μου ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ των ΚΑΠΣ και των ποσοστώσεων. Θα πρέπει να μου το πείτε επακριβώς για να το καταλάβω. Σε σχέση με τις συμβάσεις, Θα ήθελα να καταγράψουμε το εξής. Υπάρχουν χώρες που δεν έχουν τηρήσει τις δεσμεύσεις του 2006, όχι στη συνοχή, αλλά στα πιο ήπια ταμεία. Τώρα ε, μιλούσαμε για ε, την ε, προθεσμία του 2009. Αυτό το γνωρίζετε πολύ καλά. Και το γνωρίζει η κυρία Υπάρχουν όμως χώρες οι οποίες δεν έχουν τηρήσει αυτές τις ε, προθεσμίες. Θα πρέπει να δούμε ποιες είναι και οι εταιρικέ υποχρεώσεις σε αυτή την περίπτωση. Γιατί η Κομισιόν είναι υποχρεωμένη να καταβάλει ένα αντίτιμο για τις χώρες που έχουν ε, υποβάλει αίτημα. Αλλά αν παρατραβάμε αυτή την ε, προθεσμία και πάμε από τον ένα χρόνο στον άλλο, στον παράλλο, τότε η δημοσιονομική κατάσταση είναι συγκεχημένη. Ποιος πληρώνει γιατί με αυτές τις συνεχείς παρατάσεις. Αυτά θα ήθελα, σε αυτά θα ήθελα απάντηση. Η Ελίζα Μπετσουρέτερε. Ευχαριστώ. Καταρχάς, Λάμπερτ, με πάρα πολύ και Κωνσταντσα. Θυμάμαι συζητήσεις εδώ στην Επιτροπή μας που είχαν πει οι πράσινοι ότι δεν θέλουν earmarking, προσημείωση. Μετά την πρώτη ανάγνωση, όμως και πισόπλατα μας το επέβαλαν χωρίς να έχουμε καμία νομοθετική δυνατότητα επιρροής. Γιατί μας πίεζαν και δεν μπορούσαμε να υποχωρήσουμε μετά την πρώτη ανάγνωση. Και είχαν ενθουσιαστεί όλες οι μεγάλες πολιτικές ομάδες για τα μέτρα. Η σημερινή πρόταση είναι πολύ καλύτερη. Δεν είναι earmarking ε, όπως έχουμε στα τρέχοντα προγράμματα και ε, ποσοστώσεις και προγράμματα με ποσά. Εδώ επικεντρωνόμαστε σε στόχους και η ευελιξία είναι πολύ μεγαλύτερη. Αφήνει τελείως το ελεύθερο στις περιφέρειες πώς θα φτάσουν στο στόχο. Τους λένε ειδού ο στόχος και φτάστε τον. Πώς θα γίνει, από ποιο δρόμο και με ποιο μέτρο δεν μας ενδιαφέρει. Είναι σχετικά ελεύθερο. Και στον κανονισμό του Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης ε, το λέει και θα πρέπει να αλλάξει και το παράρτημα. Συμφωνώ για τους στόχους. Η προσέγγιση αυτή είναι πολύ καλύτερη και πάρα πάρα πολύ μεγαλύτερη ευελιξία και λύνει τα χέρια των περιφερειών σε σχέση με τα σήμερα ισχύοντα που ε, αναφέρονται μέτρα. Αυτό το θετικό. Και με πραγματικά εκείνοι που ήταν τόσο πολύ υπέρ των μέτρων στο παρελθόν τώρα έχουν στραφεί εναντίον τους. Νομίζω ότι αυτή η επικέντρωση στους συγκεκριμένους στόχους σε περιφέρειες που τελικά έχουν πάρα πολύ λίγα χρήματα ε, είναι πρόβλημα. Δεν μπορεί κανείς να σπέρνει δεξιά και αριστερά τα κονδύλια και μετά δεν ξέρει τι γίνονται οι περιφέρειες που έχουν πολύ μεγάλες ανάγκες, που χρειάζονται συνοχή, ε, έχουν περιορισμένους στόχους αρκετά μετριοπαθείς. Ενώ οι περιφέρειες που ε, έχει πολύ μεγάλη σημασία η τότε έχουμε μεγάλους στόχους. Αυτό με τις υποδομές δεν έχει καμία σχέση η ενέργεια, δεν έχεις δίκιο, η ενέργεια δεν μπαίνει μέσα, ε, ε, υπάρχει εξαίρεση ακριβώς για να συμβεί αυτό που χρειάζεται στο στόχο 4. Γι' αυτό βεβαίω χρειάζονται οι ενεργειακές υποδομές, αλλά εκεί έχει εξαιρεθεί. Αν κοιτάξετε τον κανονισμό, είναι πάρα πολύ συνεκτικά και με συνέπεια διατυπωμένος και το θεωρώ και σωστό. Εξαιρείται η ενέργεια. Επίσης υπάρχει πρόβλημα και ισχύει ε, στις συμβάσεις εταιρικέ σχέσεις στο άρθρο 13 και 14 αν το διαβάσει κανείς έτσι φευγαλέα θεωρεί ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαπραγματεύεται μόνο με τα κράτη-μέλη και αφήνει απ' έξω τις περιφέρειες. Η δυσκολία στο κείμενο ποια είναι. Η πολυεπίπεδη διακυβέρνηση είναι πολύ περισσότερα από αυτά που γράφονται εδώ και στο 13 και 14 δεν είναι σαφής ή αρκετά σαφής η σχέση τους και μπορεί να αλλάξει η διατύπωση. Γιατί τα κράτη-μέλη έχουν τη διακριτική ευχαίρεια να καταρτήσουν αυτή την εταιρική σύμβαση, αλλά δεν φαντάζομαι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τελικά με τις μεμονωμένες περιφέρειες να έρχεται να διαπραγματεύεται. Αυτό είναι θέμα κρατών μελών. Κάθε χώρα έχει ένα σύνταγμα, έχει έναν τρόπο διακυβέρνηση. θα πρέπει να βρει έναν τρόπο ε, συνεργασίας να προσθέσουμε μια πρόταση ε, στο 13 για το πώς θα καταρτίζονται αυτές οι συμβάσεις για να λυθεί το πρόβλημα. Ε, βέβαια πρόβλημα έχουν οι χώρες που έχουν σήμερα πολύ επίπεδη διακυβέρνηση. Στο 14 αν δούμε και διαβάσουμε με προσοχή την ουσία και το περιεχόμενο της σύμβασης το καταλαβαίνουμε, αλλά δεν είναι πάρα πολύ εύκολο να το αντιληφθεί κανείς και θα μπορούσαν τα κράτη-μέλη να το παρακάμψουν ή το παραβλέψουν, γιατί ε, είναι προϋπόθεση να υπάρχει πολυεπίπεδη διακυβέρνηση για την εταιρική σχέση. Μα έχουμε παράλληλες διαδικασίες, παράλληλα νομοθετική διαδικασία και προετοιμασίες. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Οι προετοιμασίες που γίνονται δεν έχουν νομοθετική βάση. Η βάση θα αποφασιστεί στο παραπέντε. Θεωρώ λοιπόν πολύ πιο ευτυχέ ω διαδικασία να κάνει ένα χειρίδιο Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Συστάσεις είναι αυτές στο κάτω-κάτω. Ε, ε, την ερμηνεία μπορεί να τη συζητήσει μαζί μας για το πώς όλα αυτά θα πρέπει να γίνουν ε, κατανοητά και αντιληπτά. Θα πρέπει επίσης να το πούμε από τώρα για να γράψουμε αυτό που είπατε και οι δυο σας ότι η πολυεπίπεδη διακυβέρνηση θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στην προετοιμασία των συμβάσεων και είναι και στο άρθρο 13. Θα πρέπει κάθε κράτος να εκκινήσει μια τέτοια διαδικασία, να προετοιμάζει τη σύμβαση, αλλά προϋπόθεση και αρχή είναι να υπάρχει μια πολυεπίπεδη διακυβέρνηση. Γίνεται λόγος για εταίρου, αλλά εντάξει, είπαμε είναι σαφές. Να λέμε ρητά πολυεπίπεδη διακυβέρνηση και όποιο δεν το πράττει δεν θα έχει σύμβαση. Με τη διαδικασία αυτή νομίζω πηγαίνουμε στη σωστή κατεύθυνση. Για τη δημογραφία ή ε, αυτό το εγκάρσιο συμπερίληψη σε όλα τα θέματα της δημοκρατικής εξέλιξης. Έχω αμφιβολίες κατά πόσο είναι στόχος και συμφωνώ ότι δεν είναι στόχος το άρθρο 9 αλλά να το πω διαφορετικά, ίσως στα αγγλικά, γιατί είναι σαφέστερη. Είναι κριτήριο επιλεξιμότητας, eligibility, η δημογραφική εξέλιξη. Δηλαδή, όταν είναι αρνητική κατάσταση σε μια περιφέρεια, προς τη μια ή την άλλη κατεύθυνση, γιατί έχουμε και τα δύο, και ε, περιφέρειες που ερημώνουν και επιφέρειες με πολύ μεγάλη είσοδο μεταναστών ή ε, πληθυσμού, ε, θα πρέπει να αποδεικνύεται η επιτυχία μιας περιφέρειας. Και, ε, λοιπόν, ε, αυτό είναι θέμα κριτηρίου επιλεξιμότητας στη δημογραφική εξέλιξη της κάθε περιφέρειας, εάν και κατά πόσο θα ενταχθεί. Και μπορεί να είναι κριτήριο στην προετοιμασία της σύμβασης η δημογραφική κατάσταση, αν υπάρχει έλλειμμα. Και όχι στόχος. Το θεωρώ λάθος να είναι στόχος. Πάμε σε λάθος κατεύθυνση. Οι στόχοι είναι κατά πολέμηση της φτώχειας, ε, του κοινωνικού αποκλεισμού. Όλα αυτά είναι στοιχεία που παίζουν ρόλο και στη δημογραφία βέβαια. Θέλουμε αηφόρες ε, μεταφορές Αλλιώς οργανώνονται οι μεταφορές και οι συγκοινωνίες σε περιφέρειες που είναι πιο ερημικές ή ε, άλλες που είναι πιο πυκνοκατοικημένες και έχουμε και αστικά προβλήματα στις δημόσιες συγκοινωνίες. Ωραία όλα αυτά, αλλά δεν είναι στόχος ε, το πρόβλημα το δημογραφικό, είναι μια προϋπόθεση, είναι ένα κριτήριο επιλεξιμότητας. Προσοχή να μην το πάμε σε λάθος κατεύθυνση. Η πράσινη είναι υπέρ αυτής της θεματικής συγκέντρωσης με τον τρόπο που προτείνεται εγώ είμαι και μέλος στην Επιτροπή Απασχόλησης και το συζητούν και εκεί. Σε μεγάλη πλειοψηφία η Επιτροπή αυτή είναι υπέρ ε, των στόχων του Κοινωνικού Ταμείου και όλες οι πολιτικές ομάδες κατά τα άλλα, όχι όλα τα μέλη, όλες οι πολιτικές ομάδες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το συζητάει ε, και το έχει συζητήσει και η Επιτροπή Απασχόλησης πολύ και το άρθρο 50 παίζει ρόλο και τι κρύβεται από πίσω. Το ποσοστό του κοινωνικού ταμείου αυτή τη στιγμή είναι πολύ χαμηλό στα κράτη-μέλη, αλλά έχει πολύ περισσότερες πλέον ε, αρμοδιότητες και ανάγκες να καλύψει. Συμφωνώ με αυτή τη διαβάθμιση που προτείνεται, έχει μεγάλο νόημα και στην Επιτροπή Απασχόλησης ε, νομίζω αυτά έχουν πλειοψηφία. Μπορούμε να κάνουμε και μια κοινή συνεδρίαση για να συζητήσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Έχω να κάνω κάποιες παρατηρήσεις, μερικές από τις οποίες αφορούν αυτές τις συμβάσεις εταιρική σχέσεις, Όπως είπε και ο κύριος Κοσέλσκι. Σύμφωνα με τις πρόσφατες διαπραγματεύσεις το έγγραφο, η σύμβαση αυτή θα πρέπει να είναι ένα έγγραφο που θα ξεκινά από τη βάση και θα στηρίζεται στις ανάγκες του, κρα, του κράτους μέλους. Αυτό είναι μια πρόσδεκτη εξέλιξη. Όμως, όταν συνομιλώ δεν είναι, γνωστές ε, οι, δεν είναι γνωστή η όρη συμμετοχή των ε, πόλεων και των κοινοτήτων και των περιφερειών για τη συμμετοχή τους, γιατί όλες ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για τη συμμετοχή τους και τη διαπραγμάτευση των συμβάσεων. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο αφορά κάτι που μέχρι τη στιγμή δεν έχει συζητηθεί την εκροή των 10 από την ε, πολιτική συνοχή στο συνδεδεμένο μέσο. Κατά την άποψή μου, αυτό το οποίο θα κάνει αυτό θα είναι να απομακρύνει τα, τους πόρους από έργα υποδομής στον τομέα των μεταφορών των κρατών μελών μπορούμε να σκεφτούμε ότι τυχόν θα υπάρξει ένα συμβιβασμό. Αν αφήσουμε τα 10 δι στην πολιτική συνοχής και χρησιμοποιήσουμε 40 δί από τον προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα μπορούσαμε να είχαμε επαρκείς πόρους και για τις δύο διαδικασίες. Αυτά όσον αφορά το CIF. Και η τελευταία μου παρατήρηση αφορά στο άρθρο 59 και πιο συγκεκριμένα την μη επιλεξιμότητα του ε, ΦΠΑ. Προσπαθώντας να απλουστεύσουμε τα πράγματα, στην ουσία κάνουμε πιο ακριβά τα διάφορα έργα. Ο ΦΠΑ δεν είναι επιλέξιμος. Αυτό αποτελεί μόνο εξαίρεση για μη επενδυτικά έργα και για φορείς που δεν υπόκειται σε ΦΠΑ. Θα ήθελα λοιπόν λόγω των, πρακ... συνθήκων να επιστρέψουμε στην ισχύουσα πρακτική, δηλαδή να είναι επιλέξιμο ο ΦΠΑ. Ευχαριστώ. Yes. Explain. European Commission will take... Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πάρει το λόγο προς το τέλος της συζήτησης. Θέλω καταρχήν να ευχαριστήσω τους εισηγητές που μας έδωσαν το πλαίσιο αυτής της συζήτησης. Υπάρχουν κάποια στοιχεία του γενικού πλαισίου που πρέπει να εξηγηθούν ή να καθοριστούν στην τελική εκδοχή. Θα ξεκινήσω με κάτι που θα έπρεπε να πω στο τέλος. Το συζητήσαμε με τους εισηγητές δηλαδή. Πότε θα το οριστικοποιήσουμε Είμαστε έτοιμοι να φτιάξουμε το σύστημα άσχετα από το πόσοι πόροι είναι διαθέσιμοι ή περιμένουμε την τελική απόφαση για τον προϋπολογισμό. Για το προγραμματισμό αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό, γιατί αν περιμένουμε μέχρι το τέλος της ε, διαπραγμάτευσης για τη δημοσιονομική πρακτική, θα χάσουμε όχι μόνο τον πρώτο, αλλά και τον δεύτερο χρόνο. Πρέπει λοιπόν να κάνουμε εδώ την πολιτική συζήτηση. και να αποφασίσουμε αν μειωθούν οι πόροι αυτό θα επηρεάσει το σύστημα ή όχι. Είναι απολύτως απαραίτητο. Δεν υπάρχει το κείμενο, αλλά το κείμενο αναφέρεται το ποσοστό που είναι το συμπέρασμα από, το, από την οροφή, το οποίο, το οποίο αποτελεί τη βάση. Είναι το 2,5 από τον κανονισμό. Και ε, έχει τη συνέπεια από τις λιγότερο αναπτυγμένες, περισσότερο αναπτυγμένες και μεταβατικές. Και πώς θα το κάνουμε, θα αποφασίσουμε και μετά θα προσθέσουμε το παράρτημα με τους αριθμούς. Δεύτερον, στο μέλλον η συζήτηση μπορεί να χωριστεί σε δύο μέρη. Πρώτον, τι πρέπει να γίνει και δεύτερον, πώς πρέπει να γίνει. Δεν θα πρέπει να, να μπλέξουμε το περιεχόμενο με τις μεθόδους. Φερρυπίν το τι ε, περιλαμβάνεται στους θεματικούς στόχους που περιλαμβάνει το γενικό, στο γενικό. Αλλά δεν μπορούμε να συζητήσουμε το γενικό χωρίς τη συνέπεια στο, ε, στο ΦΕΟΚΑ και στο Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης κλπ. Και όλα αυτά επηρεάζουν τις προτεραιότητες των επενδύσεων που είναι στο Περιφερειακό Ταμείο ε, Περιφερειακής Ανάπτυξης και στο ESF οι θεματικοί στόχοι επηρεάζουν επίσης το ring fencing και το λεγόμενο earmarking. Υπάρχει το earmarking, το περίφημο που αφορά τους τρεις θεματικούς στόχους, αλλά αυτή είναι η θεματική συγκέντρωση στο Ταμείο ανάπτυξη, αλλά υπάρχει ακόμα μεγαλύτερη στο ESF, γιατί η πρόταση εδώ πάει πολύ βαθύτερα. Υπάρχει earmarking εντός του ESF Δηλαδή δεν πάμε σε εθνικό επίπεδο, αλλά παραθέτω το άρθρο 4 του ESF, το earmarking πηγαίνει στο επιχειρησιακό πρόγραμμα. Άρα οι συνέπειες της έγκρισης των θεματικών στόχων είναι προτεραιότητες των επενδύσεων και δεύτερον το earmarking και τρίτον οι δείκτες. Δεν θα πρέπει λοιπόν, ε, υπάρχουν όλα αυτά τα στοιχεία της αλυσίδας. Άρα το ερώτημα είναι θα εγκρίνουμε τον κατάλογο των θεματικών στόχων και τι επιπτώσεις θα έχουν αυτοί. Δεν θα πρέπει επίσης να μας διαφεύγει ότι ο Επίτροπος Απασχόλησης δηλώνει ότι θα επικεντρωθούν σε τέσσερις θεματικούς ε, στόχους, ενώ ο Επίτροπος ε, Περιφερειακής Ανάπτυξης αναφέρει 11. Άρα στο ένα ταμείο θα, έχουμε, επικεντρωθούμε σε 11 στόχους και στο άλλο για 4 στόχους. Και όταν τεθεί το θέμα του earmarking, το θέμα του, ε, ε, για μένα τον εισηγητή είναι το earmarking είναι το 80%, το 20% κλπ. Αυτή είναι η συνέπεια. Δεύτερο στοιχείο, τα, οι συμβάσεις εταιρικής σχέσης. Σχεδόν όλα έχουν υποθεί. Όμως πρέπει να πω ότι Ίσως η δήλωση των, των πολιτικών δεν είναι σημαντική για μας. Την προηγούμενη συνεδρίαση με τους δήμαρχες, ο πρόεδρος της Επιτροπής είπε ότι θα υπάρχει εταιρική, εταιρική σύμβαση μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών. Άρα οι δήμαρχοι που ήταν εκεί ανακάλυψαν ότι οι συμβάσει θα συναυτούν μεταξύ Επιτροπής και κράτους μέλους. Στο κείμενο βλέπουμε ότι αυτό είναι ένα εσωτερικό εθνικό έγγραφο που στηρίζεται στην πολυεπίπεδη διακυβέρνηση. Σε κάποια από τα σχόλια του κανονισμού βλέπουμε ότι η σύμβαση μεταξύ σύμβαση, ε, κυβέρνησης ε, και, ε, και Ευρωπαϊκής Επιτροπής πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Το θέμα είναι μεταξύ ποιον θα είναι η σύμβαση. Και είναι προφανές. Τι σημαίνει ακριβώς ότι η σύμβαση θα εγκρίνει την ε, σύμβαση μεταξύ του εθνικού και του τοπικού. Και όσον αφορά τον κώδικα δεοντολογίας, γιατί και εδώ υπάρχει πρόταση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρουσιάσει ένα κώδικα δεοντολογίας για το πώς θα συνταχθούν οι συμβάσει εταιρικής σχέσης. Το ερώτημα είναι, είναι πιθανόν να δημιουργηθούν κώδικες διοντολογία με για 27 κράτη-μέλη με διαφορετικά επίπεδα. Εν πάση περιπτώσει το ερώτημα είναι πρέπει να υπάρχει ή δεν πρέπει να υπάρχει κώδικα. θεοντολογία. Δηλαδή στη σύμβαση εταιρική σχέσης δεν συζητάμε μόνο τη μέθοδο αλλά και το περιεχόμενο γιατί στι συμβάσει υπάρχουν ε, συμβάσει από διαφορετικά ε, ταμεία και επίσης του περίφημου τους καταλόγους πόλεων που υπάρχει το ERDF. Έτσι λοιπόν αυτό πρέπει να ε, ξεκαθαριστεί όχι για μας αλλά για αυτούς που θα υποβάλουν τις αιτήσει. Αυτοί περιμένουν και θέλουν να αρχίσουν με τις κυβερνήσεις τους να προετοιμάζουν αυτές τις ε, συμβάσεις και θέλουν να μάθουν ποια είναι η τελική εκδοχή όλο αυτού. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό το πώς αντιλαμβανόμαστε την ε, θεματική συγκέντρωση και τη σύμβαση. Και το επόμενο ερώτημα είναι πώς, ποια θα είναι η μέθοδος που θα χρησιμοποιηθεί. Και υπάρχουν πολλά νέα μέσα στον γενικό κανονισμό που ε, επηρεάζουν το ESF, αλλά είναι σοβαρό, αλλά όχι εύκολο να γίνει αντιληπτό. Τα μέσα, τα όργανα αφορούν την προετοιμασία του συστήματος υλοποίηση, το επιχειρησιακό πρόγραμμα, το θέμα της διαπίστευσης της ε, ε, της συγχρηματοδότησης και των ε, δημοσιονομικών διορθώσεων που είναι σημαντικό για μας πώς θα λειτουργήσουν αυτές και επίσης υπάρχουν και άλλα ενδιαφέροντα στοιχεία όπως ε, τοπικές ομάδες από το leader Έχουμε το κοινό σχέδιο δράσης που είναι κάτι το νέο. Υπάρχει το ITI που είναι το νέο μέσο ε, που θα χρησιμοποιηθεί και που επηρεάζει το, Ευρωπαϊκό το Περιφερειακό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και άρα πρέπει οι νέες μέθοδοι να συμπεριληφθούν στα ερωτήματα. Πρέπει με, το, με τα νέα μέσα να μάθουμε ποιο μέσο θα χρησιμοποιηθεί για ποιο σκοπό, γιατί δεν μπορούν όλα να χρησιμοποιηθούν για όλους τους σκοπούς. Πρέπει να είναι ξεκάθαρο ποιε είναι οι συνέπειε τη όλη αυτή τη προσπάθεια. Εν πάση περιπτώσει, πολλά μένουν ακόμα να γίνουν και αυτή τη φορά ο Γενικό Κανονισμό συμπεριλαμβάνει πάρα πολλά στοιχεία του υπολείπου κανονισμού και άρα δεν μπορούμε να λύσουμε το πρόβλημα στον συγκεκριμένο κανονισμό αν δεν είναι ξεκάθαρη η θέση του γενικού. Άρα πρέπει να συνεργαστούμε. Δεν μπορούμε να δουλέψουμε χωριστά γιατί θα είναι παράλογο, δεν θα είναι λογικό να το κάνουμε αυτό. Επαναλαμβάνω, έχουμε το πλαίσιο αλλά πρέπει να γίνουμε πολύ καλή δουλειά για να ξεκαθαρίσουμε όλα τα στοιχεία που είναι πολύ ενδιαφέροντα αλλά και πάρα πολύ σύνθετα. Ευχαριστώ. Βίκτορ Μποστινάρα, παρακαλώ. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε, πολύ. Τα περισσότερα προβλήματα ήδη αναφέρθηκαν. Θα ήθελα εγώ μόνο να παραπέμψω στα εξής. Συμφωνώ και εγώ και η εταιρική σύμβαση δεν θα πρέπει να είναι ένα διμερές έγγραφο μεταξύ Ευρωπαϊκής Επιτροπής και κράτους μέλους. Αυτό δεν είναι πολυεπίπεδο συμβόλαιο, ούτε πολυεπίπεδη διακυβέρνηση όταν δεν υπάρχει χώρος και δυνατότητα ε, λόγου για το τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Θα πρέπει να είναι κάτι που να ορίζει σαφώς το ρόλο σου και τη σημασία των περιφερειακών και των τοπικών φορέων για τις θεματικές προτεραιότητες θα ενθάρρυνα πάρα πολύ την ιδέα που λέγει ότι στη διαπραγμάτευση με τα κράτη-μέλη, τα κράτη θα έχουν περισσότερη ευελιξία, διακριτική ευχέρεια για να εφαρμόζουν και να προσαρμόζουν στη δική τους πραγματικότητα και στις δικές τους ανάγκες σημαντικές προτεραιότητες. Γιατί διαφέρει πάρα πολύ η κατάσταση από χώρα σε χώρα για την ευελιξία και τις ποσοστώσεις και πάλι θέλω περισσότερο χώρο για διαπραγμάτευση από την πλευρά των κρατών μελών. Γιατί καμιά φορά είναι τεράστιες οι διαφορές και οι ιδιαιτερότητες των χωρών. Και αυτή η περιχαράκωση, το ring fencing, ε, θα ήθελα να προτείνω την εξή ιδέα, να διαπραγματεύονται τα κράτη-μέλη με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πάντα έχοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες τη κάθε χώρας για το κοινωνικό στρατηγικό πλαίσιο. Θα πρέπει το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο να εγκρίνει αυτά και όχι μέσω κατεξουσιοδότηση πράξεων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να θεωρείται κάπως ως παράρτημα στο γενικό κανονισμό και όχι κάτι που ανήκει ε, σε μια διαφορετική νομοθεσία. Γιατί αυτό θα δώσει και μεγαλύτερη προβολή και ορατότητα όταν είναι νομοθέτημα και όχι κατεξουσιοδότηση πράξη. Και επίσης θα δείξει και τι σημασία έχει το έγγραφο. Έχει άλλο ειδικό βάρος όταν εγκρίνεται από το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο. Διαφωνώ κάθετα, και όχι εγώ προσωπικά, μιλάω εξ ονόματος πολιτικής μου ομάδας. Και συναντηθήκαμε και τους σκιώδης είτε στην περασμένη εβδομάδα. Είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι η μακροοικονομική αιρεσιμότητα δεν θα πρέπει να θεωρείται τμήμα του γενικού κανονισμού Για οποιονδήποτε κανόνων που διέπουν τα ταμεία συνοχής. Διότι αυτός θα είναι ένας νέος τρόπος να πλήττονται οι κοινότητες που έχουν προβλήματα. Θυμάστε πριν από δύο εβδομάδες τι συμφώνησε το Συμβούλιο. Η λεγόμενη Δημοσιονομική Ένωση θα έχει μεγάλο αντίκτυπο, για να μην πω δραματικό, στη δυνατότητα που θα έχουν τα κράτη-μέλη όχι μόνο να ασκούν οικονομικές πολιτικές, αλλά και να συγχρηματοδοτούν τις κοινοτικέ πολιτικές. Και αν έρθουν επιπλέον κυρώσει, ε, δεν θα μπορέσουν καθόλου να αξιοποιήσουν αυτή τη δυνατότητα. Διαφωνώ ριζικά με την ιδέα αυτή της μακροοικονομικής αιρεσιμότητας και σταθερότητας ως ε, ένα από τα κριτήρια. Και υπάρχουν και άλλα στοιχεία που έχουν σχέση περισσότερο με τη δική μου γνωμοδότηση, αλλά αυτό δεν είναι του παρόντος. Ευχαριστώ. Very much. Manner. Ευχαριστώ. Λέει η κυρία Μάνερ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συνεισηγητές για αυτό το εξαιρετικό έγγραφο σε σχέση με αυτό τον κανονισμό. Πολλά ακούστηκαν και νομίζω ότι έχουν καλυφθεί πολλά. Ως προς τα τέσσερα σημεία, νομίζω ότι μπορώ να υποστηρίξω τους εισηγητές και αυτά που είπε ήδη η Κωνσταντσε Κρέλ στα εισαγωγικά της σχόλια σε σχέση με την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση Συμφωνώ με αυτά που είπε ο προηγούμενος ομιλητής. Νομίζω ότι μπορούμε να φτάσουμε σε μία συνεργασία σε περιφερειακό και άλλα επίπεδα ως προς τις εταιρικέ συμβάσεις και την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση. Σύμφωνα με αυτά που ήδη ελέγχθησαν, ως προς τις θεματικές προτεραιότητες χρειαζόμαστε ε, ευελιξία, όπως είπε και η Κωνσταντσε Κρέλ. Νομίζω ότι θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε καλύτερα τα ταμεία και για έργα υποδομής και προγράμματα υποδομής και πιστεύω ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα ταμεία για προγράμματα ε, διεθνικά. Γιατί πολλές φορές έχουν μεγάλη σημασία για ιδιαίτερες, ε, για συγκεκριμένες περιφέρειες. Ως προς την ευελιξία βεβαίως θα πρέπει να υπάρχει ένα συγκεκριμένο εύρος, ως προς την αντιστήχηση, το earmarking, ε, εδώ έχω ορισμένε επιφυλάξεις, θα πρέπει να ακούσουμε τις περιφέρειες καταρχήν. Κωνσταντσε ε, μίλησε και για δημογραφικές καθαρά προτεραιότητες. Εδώ θα πρέπει να κινηθούμε με βάση τον γενικό κανονισμό. Βεβαίως, οπωσδήποτε η γύρανση του πληθυσμού αποτελεί μια μεγάλη πρόκληση για μας, ε, για το μέλλον και θα πρέπει να ληφθεί υπόψη από τον γενικό κανονισμό. ως προς τις εδαφικές, ε, το, την εδαφική διάσταση νομίζω ότι ε, αυτή η συζήτηση θα συνεχιστεί στο μέλλον. Ο Γιακή έχει φύγει, η επόμενη ομιλήτρια. Ευχαριστώ Πρόεδρε, λέει η κυρία Πέρες, ε, σας ευχαριστώ Και θα ήθελα να πω ότι οι προλαλήσοντες ε, με οδήγησαν στο να καταλάβω πολλά από τα ζητήματα αυτά σε σχέση με τις ε, ε, επενδύσεις. Νομίζω ότι εδώ εφήγησαν αρκετά ζητήματα. Θα επικεντρωθώ σε ζητήματα αρχής, γιατί νομίζω ότι ότι ο νομοθέτης, δηλαδή εμείς, θα πρέπει να βρούμε τον καλύτερο τρόπο χρήσης των ταμείων. Ως προς την ευελιξία ήδη μιλήσαμε αρκετές φορές για την ευελιξία να βρούμε την καλύτερη αποτελεσματικότητα αυτών των μέσων και γι' αυτό θα πρέπει να δούμε τις εθνικές και περιφερειακές ιδιαιτερότητες θα πρέπει να εισακουστούν οι περιφέρειες γιατί γνωρίζουν καλύτερα για την χρήση των κονδύλιων. Έχω ορισμένε αμφιβολίες ως προς τους, ε, τα όρια που προτείνει η Επιτροπή ιδιαίτερα ως προς το ΕΚΤ. Και ως προς την αρχή της απλούστευσης, θεωρώ ότι η πρόταση της Κομισιόν ε, είναι ελληματική ως προς ουσιαστικά στοιχεία απλούστευσης και νομίζω ότι δεν μπορεί να γίνει πλήρης απορρόφηση των κονδυλίων διότι δεν υπάρχει μία σωστή πολιτική συνοχή. Όπως είπε και ο Μποστινάρου, θα πρέπει να άρουμε την μακροαιρεσιμότητα και εξάντε και εξπόστ. Σε σχέση με τις εταιρικές συμβάσεις, συμφωνώ με αυτά που είπαν οι εισηγητές και η Επιτροπή ότι θα πρέπει να έχουμε μια πολυεπίπεδη διακυβέρνηση. Επειδή όμως θέλουμε να είμαστε αποτελεσματικοί θα πρέπει να έχουμε και πρακτικό καθαρά πνεύμα και προσέγγιση ως προς τα διάφορα επίπεδα διακυβέρνησης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ ε, Φραντσέσκο Ντάντζελης. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω καταρχήν τους εισηγητές για την εξαιρετική αυτή εργασία και να εκφράσω ορισμένες σκέψεις εντάχει. Ως προς τις ε, γενικές, ε, το γενικό πλαίσιο και ως προς την πρόταση της Επιτροπής δεν θεωρώ ότι θα πρέπει να ορίσουμε την πολιτική συνοχής με βάση το σύμφωνο σταθερότητας και ανάπτυξης. Εάν την υπαγάγουμε στο σύμφωνο, τότε δεν λαμβάνουμε υπόψη τις ε, γενικότερες πολιτικές που μας ενέπνευσαν ως προς την πολιτική συνοχής, ως προς τα γενικότερα σχόλια. Μιλάμε για έναν κανονισμό συμπεριληπτικό και νομίζω ότι χρειάζεται για την καλή διαχείριση του πλαισίου. Επειδή γίνεται όμως λόγος για το γενικό πρόγραμμα έρευνας που θα ενταχθεί στο στρατηγικό πρόγραμμα, και την έρευνα και την ανάπτυξη θα τη δούμε ξεχωριστά από την καινοτομία, θα πρέπει να δούμε εάν υπάρχει συνάφεια μεταξύ των δύο. Στα πλαίσια τώρα των συμφωνιών, των συμβάσεων εταιρικής σχέσης, επειδή ε, οι προσυπογράφοντες είναι οι περιφέρειες, θα πρέπει να δούμε πώς θα ισχύσει η αρχή της επικουρικότητας διότι οι περιφερειακοί φορείς θα πρέπει να συμμετέχουν άμεσα και να δούμε ποιοι θα είναι και οι επικεφαλής αυτής της διαδικασίας. Δηλαδή, οι περιφέρειες διαχειρίζονται την πολιτική συνοχής επί της ουσίας. Τέταρτον, ως προς τις εταιρικές συμβάσεις, συμβάσεις εταιρικής σχέσης, θα πρέπει να τις εντάξουμε μέσα στα λειτουργικά προγράμματα. Και μέσα στα πλαίσια της αιρεσιμότητας θα πρέπει να ορίσουμε και γενικότερα ζητήματα αρχής. Ως προς την ευελιξία και τις ποσοστώσεις, θεωρώ ότι οι θεματικές προτεραιότητες εντάσσονται στην στρατηγική 2020. Συμφωνώ όμως, όπως είπαν και οι δύο εισηγητές, ότι δεν υπάρχει κατάλληλη ευελιξία έτσι ώστε να λάβουμε υπόψη συγκεκριμένες προαπαιτήσεις περιφερειακής ανάπτυξης και χρειάζονται έρευνες για τις υποδομές, έργα υποδομής ιδιαίτερα στα νέα κράτη-μέλη. Ως προς τις ποσοστώσεις δεν θα πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένες αριθμητικές καθαρά ποσοστώσεις και να λάβουμε υπόψη και την κοινωνική διάσταση της πολιτικής συνοχής ως προς την απλούστευση τη θεωρώ ύψης της σημασίας διότι μιλάμε για την πρόσβαση και για την ευχέρεια της χρήσης των πόρων. Αυτό είναι ένα θέμα που οδηγεί σε δυσχέρειες και που πρέπει να διευθετήσουμε. Θα πρέπει να υπάρχει καλύτερη προσβασιμότητα στην χρήση αυτή, στους πόρους αυτούς. Και νομίζω ότι η πρόταση της Επιτροπής δεν κινείται προς αυτή την κατεύθυνση. Ερμήνια Ματσάν. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι η αρχική ιδέα της Επιτροπής για έναν ενιαίο κανονισμό για όλα τα ταμεία προωθεί την απλούστευση αυτή και συμφωνώ με τους ε, προλαλήσαντες και ιδιαίτερα με τον κύριο Ντεάντζελης γιατί η Επιτροπή δεν έχει φτάσει, δεν ανταποκρίνεται σε αυτό το στόχο, δεν επιλύονται τα προβλήματα διαχείρισης με μία απλούστευση και μόνο. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να καταβάλουμε μεγαλύτερες προσπάθειες, άλλου είδους προσπάθειες, ως προς την καλύτερη και μεγαλύτερη χρήση των ταμείων που διέπει αυτή την οργάνωση των κανονισμών έχει αδυναμίες. Και ο κύριος Γκούτμαν μίλησε για την απλούστευση και να υπάρχει μια μεγαλύτερη ευελιξία μεταξύ ταμείων έτσι ώστε να υπάρχει ένας ρυθμιστικός μηχανισμός για μεγαλύτερη ευελιξία μέσα σε κάθε ταμείο. Θα πρέπει να κατανοήσουμε τι αλληλεπίδραση υπάρχει μεταξύ ταμείων και κατά πόσο μπορούμε να φτάσουμε σε μια άλλη συμπληρωματικότητα. Ιδιαίτερα ως προς το Ταμείο Συνοχής που έχει έναν εξορισμό, περιορισμό. Θα πρέπει να κατανοήσουμε πώς μπορούμε να κινηθούμε και πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα άλλα ταμεία έτσι ώστε να ορίσουμε το συμπληρωματικό χαρακτήρα που υπάρχει στα διάφορα ταμεία ε, μέσα στα πλαίσια της στρατηγικής 2020. Ως προς τις εταιρικέ συμβάσεις, συμφωνώ με όλους τους προλαλήσαντες ότι χρειάζονται περισσότερες διασαφήσεις. Δηλαδή, από το γενικό ρυθμιστικό πλαίσιο Πολλά ζητήματα δεν είναι σαφή ως προς την ε, συμμετοχή, δημοκρατική συμμετοχή των τοπικών αρχών. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει μια ευαισθητοποίηση και μια μεγαλύτερη ευθύνη όλων των φορέων. Όλα αυτά θα πρέπει να ενταχθούν στις περαιτέρω διευκρινήσεις του κανονισμού. Θα πρέπει να δούμε πώς ορίζονται και αυτές οι συμβάσεις, όπως είπε και ο συνάδελφος Μποστινάρου. Διότι όλα αυτά ξεκινούν από τις περιφέρειες και όχι από τα κράτη-μέλη. Ως προς την μακροερεσιμότητα, διαφωνώ κι εγώ, θα ήθελα όμως να μας διευκρινίσει η Επίτροπη κατά πόσο αυτές οι μακροοικονομικές προβλέψεις συνάδουν με την ε, πολιτική συνοχής. Γιατί δεν φαίνεται να υπάρχει ένας τέτοιος συνεκτικός κρίκος. Θα κρατήσει αυτή τη θέση της Επιτροπή. Γιατί διαφορετικά φαίνεται ότι έχουμε να κάνουμε με ένα πλαίσιο κυρώσεων το οποίο δεν μπορεί να ενταχθεί στην ε, πολιτική συνοχής. Βεβαίως θα υπάρχουν μεγαλύτεροι έλεγχοι, σοβαρές κυρώσεις, γιατί όπως είδαμε από τον προγραμματισμό μας τα πράγματα δεν ε, εξελίχθηκαν καλά. Δεν μπορούμε όμως αυτό να το εντάξουμε στους μακροοικονομικούς δείκτες, διότι αυτό αποτελεί αρνητική κύρωση κατά της πολιτικής συνοχής. Τώρα, ως προς τις περιφέρειες, δεν ξέρω κατά πόσο εισαγωγή νέων περιφερειών δεν θα οδηγήσει σε όλισθήσει σπόρων από μία κατηγορία σε άλλη. Και πέρα από τις ε, κυρώσεις και τη σύρρυκνωση των πόρων, στην ουσία πλήττει τις περιφέρειες που βρίσκονται μέσα στους συγκεκριμένους στόχους και ιδιαίτερα το στόχο 1. Πρόκειται για ένα ποσό που είναι ήδη μικρότερο. Αν, μπει και άλλοι, αν μπουν και άλλες περιφέρειες, τότε θα έχουμε νέες κατηγορίες οι οποίες θα έχουν επιπτώσεις επί των ήδη περιορισμένων πόρων. Πώς θα επαναδιοργανώσουμε τους στόχους και πώς θα ενταχθούν και άλλες περιφέρειες συρρυκνώνοντας τους πόρους. Τέλος, ως προς το Ταμείο για τις υποδομές μέσα στα πλαίσια του Ταμείου Συνοχής, νομίζω ότι η πρωτοβουλία της Επιτροπής είναι πολύ καλή, αλλά υπάρχουν επικρίσεις. διότι δεν υπάρχει δυνατότητα αυτόνομης διαχείρισης από τις περιφέρειες. Δηλαδή, αυτά τα δέκα δις πώς θα απορροφηθούν. Θα απορροφηθούν από επίπεδο κεντρικών κυβερνήσεων. Αυτό δεν είναι σωστό. Επίσης, ποια κριτήρια θα χρησιμοποιηθούν για να εξατομικεύσουμε τις προτεραιότητες που δεν ορίζονται από την ίδια την πρόταση της Κομισιόν, διότι ως προς το Ταμείο Συνοχής, και αυτό είναι το καινοτόμο στοιχείο, χρειάζεται μια διασάφηση από πλευράς Επιτροπής για να μην γίνουν στρεβλώσεις. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πριν δώσω το λόγο στο Γενικό Διευθυντή, θέλω να πω το εξή. Αντιλαμβάνομαι ότι όλοι ανησυχούμε για ένα θέμα, πολλά, για πολλά, αλλά ένα που κατέστη απόλυτα σαφές σήμερα είναι να φροντίσουμε ότι οι κανονισμοί να δημιουργήσουν τις συνθήκες να συμμετέχουν, να εμπλακούν και οι περιφέρειες. Και άρα δεν θα πρέπει πιστεύω να κοιτάμε μόνο ακριβώς το περιεχόμενο του ε, κανονισμού, δηλαδή τη σύμβαση εταιρικής σχέση που εμπλέκει τις αρχές, αλλά πρέπει να δούμε και όλες τις άλλες λύσεις από τη σκοπιά του εάν και κατά πόσον διευκολύνουν την συμμετοχή των περιφερειών. Ας πούμε, αν ε, είναι, στοχευμένο, ε, προ προς τα αποτελέσματα, σημαίνει ίσως ότι πρέπει να βρούμε ε, δείκτες που δεν μπορούν να εντοπιστούν σε μικρότερες περιφέρειες κλπ. Είναι πολλά πράγματα που μπορούν να δυσκολέψουν ε, και να κάνουν δύσκολο για τις, τις περιφέρειες να συμμετάσχουν και ως εκ τούτου να υπονομεύσουν την ε, προθυμία τους να κινηθούν περισσότερο στο πλαίσιο των περιφερειακών προγραμμάτων. Τώρα θα δώσω το λόγο στον Νίκολας Μάρτιν, ο οποίος ε, θα ήθελα να θίξει κάποια θέματα. Αλλά πριν το κάνω αυτό, ο Έρικ έφυγε, αλλά είχε παραμείνει εδώ, στο πρώτο μέρος της συνεδρίασης. Ήταν ε, ο σύνδεσμός μας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Γενικής Διεύθυνσης. Η Γραμματεία συνεργάστηκε πολύ καλά μαζί του. Θα θέλαμε να τον ευχαριστήσει γιατί αυτή ήταν η τελευταία του συνεδρίαση. Σας παρακαλώ να του διαβιβάσετε τα σχόλιά μου και να δούμε ποιος θα αποφασίσετε να είναι ο επόμενος σύνδεσμος. Θα τους υποδεχτούμε με μεγάλη χαρά. Λοιπόν, Νίκολας Μάρτιν, έχεις το λόγο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Βεβαίως και θα διαβιβάσω αυτά που είπατε στον ε, Ερικ. Όπως ξέρετε θα παραμείνει στην Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής και άρα θα έχετε τη δυνατότητα να τον έχετε στην ε, ε, Επιτροπή σας ως Διευθυντή. Και μόλις οριστεί ο αντικαταστάτης του θα σας ειδοποιήσουμε. Θεωρούμε ότι αυτό είναι ένα από τα βασικά έργα του υπεύθυνου συνδέσιμου της Επιτροπής. Είναι πολύ, σημαντικ... Ε, πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά τα εκτεταμένα και διαφορετικά σχόλια. Έχουμε ένα μακρύ κατάλογο σημείων, υπάρχουν όμως κάποια τα οποία είναι κρίσιμες σημασίες και θα μου δοθεί ευκαιρία να επανέλθω και να ξεκαθαρίσω, να δώσω τη σκοπιά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε κάποια από αυτά. Όταν ε, πήρα το λόγο νωρίτερα, κάποια από τα σημεία που προέκυψαν από τη συζήτηση στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων ε, είπα ότι ξαναπροέκυψαν ε, και σήμερα το κοινό πλαίσιο στρατηγικής είναι ένα από αυτά. Θα ήθελα ίσως να εξηγήσω ποιος είναι για μας ο κρίσιμος ρόλος του κοινού στρατηγικού πλαισίου. Φυσικά θεωρούμε ότι είναι ένα στρατηγικό έγγραφο, ένα εξορισμού σημαντικό έγγραφο από τη σκοπιά αυτή. Όμως ένα έγγραφο που πρέπει να έχει αξία για τα κράτη-μέλη. Ιδάλλως μπορεί απλώς να είναι ένα υψηλού επίπεδου κείμενο που δεν θα βοηθάει όμως τα κράτη-μέλη τα οποία θα ξεκινούν την όλη διαδικασία προετοιμασίας των προγραμμάτων της επόμενης περίοδου. Θέλουμε να φροντίσουμε να επιτευχθεί αυτό που ε, στο οποίο στοχεύουμε. Την ε, ιδέα της ε, ολοκλήρωσης των ταμείων αυτών, της χρήσης τους για την πολιτική συνοχής και για την ενεργοδοτική ανάπτυξη και την αλληλεία κλπ. Και να μπορέσουμε να κάνουμε σωστή διάρθρωση ανάμεσα στη θεματική προσέγγιση και την εδαφική προσέγγιση η οποία αναφέρθηκε από πολλούς ομιλητές σήμερα. Είναι ένα θέμα που και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή την απασχολεί και ε, βλέπουμε ότι η, ε, ε, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, είναι, το, το, το CSF είναι ένα σημαντικό στοιχείο. Πρέπει λοιπόν να δούμε ποιο είναι, τι πρέπει να περιλαμβάνει το CSF κατά την άποψη της Επιτροπής, να έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε το έγγραφο αυτό. Εδώ σε αυτό το κοινοβούλιο θα ακούσετε αν έχουμε κοινή προσέγγιση για το τι μπορεί να κάνει αυτό το CSF, το κοινό στρατηγικό πλαίσιο. Και αυτό θα μας βοηθήσει να προχωρήσουμε ε, στο ε, θέμα της διαδικασίας. Ίσως ε, ε, συμφωνώ με αυτό που είπε ο κ. Ε, Διάντζελης ε, στη σχέση με τον ορίζοντα του 2020. Είναι ένα βασικό θέμα, αλλά και με άλλες πολιτικές, εκτός της πολιτικής συνοχής, διότι αυτό είναι ένας από τους βασικούς στόχου να ενσωματωθούν εκεί, να υπάρξει μια ολοκλήρωση όλων των πηγών χρηματοδότηση. Συμφωνώ, όπως είπε η κυρία Κρέρ, ότι υπάρχει μια σχέση. Το CSF ε, σχετίζεται με την θεματική συγκέντρωση, με τις ε, συμβάσει. Αναγκαστικά αλληλεπιδρούν όλα αυτά και πολλοί από του ομιλητέ σήμερα ασχολήθηκαν με τη Σύμβαση Εταιρική σχέση που πολύ σωστά θεωρείται κρίσιμη σημασία γιατί προσφέρει στο κράτος μέλος την γενική εικόνα του πώ θα χρησιμοποιηθούν οι πόροι και από εκεί και πέρα το βασικό είναι τα, η πολυεπίπεδη διακυβέρνηση. Είναι ενδιαφέρον που ε, ε ακούμε και συγκρίνουμε τις ανησυχίες που ακούγονται εδώ με αυτές που ακούγονται στο Συμβούλιο. Αυτό που έχει επιδιώξει με την πρότασή της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι να εξισορροπήσει δύο ειδών ανησυχίες. Ανησυχίες που ακούγονται στο Συμβούλιο. Αυτές έχουν κυρίως σχέση με το σεβασμό προς το ε, θεσμικό πλαίσιο που έχει δημιουργηθεί, την πολυμορφία των θεσμικών ρυθμίσεων και τις διαφορές που μπορεί να προκύψουν στα ομόσποδα κράτη-μέλη και τα θέματα που αφορούν κράτη-μέλη με περισσότερο συγκεντρωτική δομή. Ε, βεβαίως υπάρχουν και εδώ ανησυχίες που ε, ε, ενδιαφέρουν να, που αφορούν το, ε, την, το να δοθεί παρκής δυνατότητα στις περιφέρειες και τους Δήμους να παίξουν τον πλήρη, τον πλήρη ρόλο τους. Είναι δύσκολη η ισορροπία εδώ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επεδίωξε να πετύχει την ισορροπία αυτή διατυπώνοντας το ρυθμιστικό πλαίσιο με τρόπο που κατά την άποψή μας επιτρέπει να ληφθεί ληφθούν υπόψη ή τα, διάφορα, τα διαφορετικά θεσμικά πλαίσια. Ταυτόχρονα όμως να δοθεί και αυτή η όθηση προς ε, μια ενισχυμένη πολυεπίπεδη διακυβέρνηση. Ο κώδικας διοντολογίας για μας είναι ένα σημαντικό στοιχείο στην όλη αυτή προσπάθεια και γι' αυτό του, ε, ε, τον ενισχύσαμε κάπως και θεωρούμε ότι είναι ένα έγγραφο που πρέπει να εγκριθεί ως κατεξουσιοδότηση πράξη. Ε, ε, θα περιλαμβάνει στοιχεία που πράγματι ε, θα ενθαρρύνουν όλα τα κρατημέλη να εξασφαλίσουν ότι θα υπάρξει επαρκής εμπλοκή όλων των ενδιαφερομένων και των περιφερειακών αρχών και δήμων. Αυτό όμως δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να ταιριάζει σε όλους. Τώρα, όσον αφορά το ποιο θα κάνει τη διαπραγμάτευση, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι στην πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπάρχει η υποβολή της σύμβασης με τα επιχειρησιακά προγράμματα σε ένα πακέτο. Το, η σύμβαση είναι το έγγραφο που καλύπτει όλα τα κρατημέλη και άρα η διαπραγμάτευση θα γίνει μεταξύ Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ε, του ε, κράτους μέλους. Όμως θεωρούμε ότι το έγγραφο αυτό είναι αναγκαστικά αποτέλεσμα εσωτερικών συζητήσεων και διαπραγματεύσεων με την συμμετοχή όλων όσοι πρέπει να εμπλακούν σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο για να ε, οδηγηθούμε στις αποφάσεις που περιλαμβάνει η σύμβαση, πώς θα χρησιμοποιηθεί η χρηματοδότηση, το είδος ε, του έργου, το είδος ε, του περιφερειακού ή των ε, εθνικών ή κεντρικού προγράμματος, η κατανομή της χρηματοδότησης, η επιλογή των θεματικών στόχων. Μια σειρά λοιπόν από κρίσιμες αποφάσεις πρέπει να ληφθούν και αυτές ανακεφαλαιώνονται την ε, Σύμβαση εταιρική Σχέσης, αλλά μπορεί να είναι μόνο αποτέλεσμα μια εντατικής συζήτησης, διαβούλευσης και ε, λήψη αποφάσεων σε εθνικό επίπεδο. Ω εκ τούτου, για τη διαπραγμάτευση, αυτό που είναι απαραίτητο είναι η σύμβαση να, διαπραγματευτεί σε εθνικό επίπεδο, να τη διαπραγματευτεί σε εθνικό επίπεδο η Επιτροπή με το κράτος μέλος, αλλά ε, πρέπει να έχει προκύψει και από συζήτηση με τις ε, ε, αρχές που εμπλέκονται στο πρόγραμμα. Είναι μια διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί μετά την υποβολή του πακέτου και η οποία θα οδηγήσει πρώτον στην έγκριση από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της Σύμβασης και, που θα, και την οποία θα ακολουθήσει η έγκριση των χωριστών προγραμμάτων. Τώρα, όσον αφορά αυτό το ζήτημα της εξισορρόπησης της θεματικής προσέγγισης με την εδαφική προσέγγιση. Ίσως λόγω αυτής της σχέσης με την Ευρώπη 2020 ε, έχουμε δει τη διατύπωση του, της θεματικής, ε, θεματικού καταλόγου και δημιουργείται η αίσθηση μιας ε, έλλειψης ισορροπίας. Ε, η δική μας πρόταση ίσως ε, δίνει υπερβολική έμφαση στο κλαδικό στοιχείο, στο δομιακό στοιχείο και δεν παίρνει υπόψη του επαρκώς το εδαφικό στοιχείο. Αυτή δεν ήταν η αρχική μας διάθεση γιατί σαφώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πιστεύει ότι η πολιτική συνοχής στηρίζεται σε μια εδαφική προσέγγιση που έχει τις ρίζες της στις συγκεκριμένες εδαφικές ανάγκες. Και αυτό είναι ενσωματωμένο στο περιεχόμενο της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης και στο πρόγραμμα. Και όπως είπα, αυτό που θέλουμε να ξεκαθαρίσουμε είναι ότι θέλουμε να υπάρχει ισορροπία ανάμεσα σε αυτό και το κοινό στρατηγικό πλαίσιο. Θεωρείτε όμως και εσείς ότι υπάρχουν στοιχεία που έχουν ε, ε, ε, συμπεριληφθεί για να αντιμετωπιστούν κάποιες συγκεκριμένες εδαφικές ανάγκες όπως η δυνατότητα να υπάρξουν ολοκληρωμένες ε, ε, χωροταξικές εδαφικές επενδύσεις και ολοκληρωμένες αστικές στρατηγικές. Όμως αυτή είναι μια διαρθρωμένη προσέγγιση και που πρέπει να προκύψει από τα επιχειρησιακά προγράμματα της συμβάσης σχέσης γιατί πρέπει από τον κανονισμό να ε, προκύψει υπάρχει εκεί η ανάλυση των ανάγκων σε ε, ε, στο εδαφικό πεδίο. Τώρα όσον αφορά τη θεματική συγκέντρωση Βεβαίω η αφετηρία εδώ είναι η συμφωνία για το, τι, για το γιατί υπάρχει ανάγκη συγκέντρωσης, υπάρχει ενισχύ της επιπτώσει των πόρων και ε, οδηγεί ε, στην επίτευξη των κοινών στόχων. Υπάρχουν μηχανισμοί όπως η το να μην, μπορούν, να μην εμποδίζονται οι σωστέ, οι, να ληφθούν υπόψη οι πραγματικές ανάγκες σε εδαφικό επίπεδο. Βεβαίω τα ταμεία λειτουργούν διαφορετικά. Το Ταμείο Συνοχή έχει μια δική του ενδογενή συγκέντρωση που προκύπτει από τη συνθήκη. Ε, το ε, ESF επικεντρώνεται σε τέσσερις ε, θεματικούς ε, άξονες, ενώ το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης έχει 11 θεματικούς στόχους. Υπάρχει λοιπόν μια λογική ε, πίσω από τους διαφορετικούς μηχανισμούς. Για να καταλήξουμε σε κάτι λειτουργικό, πρέπει να γίνουν επιλογές σε κάποιες περιπτώσεις και μάλιστα δύσκολες, ε, να ληφθούν δύσκολες αποφάσεις. Η φύση του μηχανισμού αποτέλεσε αντικείμενο μακρά σκέψης και τελικά η άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ήταν «Ε, αν δεν έχουμε συγκεκριμένα ποσοστά, συγκεκριμένα σημεία αναφοράς δεν θα λειτουργήσει, δεν θα στηθεί αυτός ο μηχανισμός. Επίσης αντιλαμβανόμαστε την ανάγκη που υπάρχει για ευελιξία. Αυτό το οποίο ίσως δεν έχει ε, γίνει ε, σοβαρά αντιληπτό είναι η ενσωματωμένη ευελιξία του Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης ε, με ποσοστό που επιτρέπει τις ε, τοπικές τις περιφερειακές ανάγκες να ληφθούν υπόψη. Δηλαδή δεν έχει κάθε περιφέρεια τις ίδιες ποσοστώσεις. Επίσης, έχουμε και μια διαφοροποίηση ανά κατηγορία επιτροπής. Οι λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες έχουν, δεν έχουν κανένα περιορισμό στον, στην επιλογή των θεματικών. Οι περιφέρειες μετάβασης το 40% και για τις πιο ανεπτυγμένες 20% χωρίς περιορισμούς. Ήδη λοιπόν γίνεται μια διαφοροποίηση. Και ένα άλλο σημαντικό σημείο που σχετίζεται και με ένα ζήτημα που ετέθη για την ευελιξία των δικαιούχων. Οι διάφορες ε, ε, εργασίες μπορούν να χρηματοδοτηθούν από διαφορετικές πηγές για το ίδιο πράγμα και αυτό επιτρέπει μια ευελιξία σε αυτό το επίπεδο. Σημαντικό. Ένα συγκεκριμένο ζήτημα, για να έρθω στα συγκεκριμένα που προέκυψαν από τη συζήτηση, στην Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία, το θέμα της διαμεθοριακής υποδομής και εδώ έχουμε ένα κοινό στόχο με την ε, Κομισιόν η οποία στο άρθρο 6 του κανονισμού ETC κάνει ανα, ρητή αναφορά στη χρήση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερικής Ανάπτυξης που θα χρησιμοποιηθεί για τα διαμεθοριακά. Αυτό ήδη έχει ληφθεί υπόψη. Τώρα, το θέμα της ε, απλούστευσης. Δεν έχω τώρα χρόνο να περιγράψω όλους τους τρόπους με τους οποίους θεωρούμε ότι έχουμε απλουστεύσει το θεσμικό πλαίσιο σε σχέση με το παρελθόν. Αποτελεί ε, ένας από τους βασικούς στόχους της πρότασης της Κομισιόν και είναι ευπρόσδεκτη η ευκαιρία να γίνει συζήτηση ε, επ' αυτού. Είναι πολύ σημαντικό ποιοι οι τρόποι. Ε, υπάρχει μεγάλος αριθμός τρόπων με τους οποίους οι κανόνες βοηθούν την ευελιξία και ε, δημιουργούν αναλογικότητα. Έχουμε κάνει ένα σημαντικό βήμα πρόοδου. Ένα παράδειγμα, το γεγονός ότι υπάρχει κοινή σειρά ε, κανόνων επιλεξιμότητας δεν είναι απλό και όσον αφορά τους δικαιούχους αυτό οπωσδήποτε ε, έχει σημασία. Από την πλευρά τώρα του οικονομικού ελέγχου έχουν ενσωματωθεί συγκεκριμένες διατάξεις, ώστε οποιοδήποτε έργο κάτω των 100.000 ευρώ μπορεί μόνο να ελεγχθεί μία φορά στη διάρκεια της περίοδου εφαρμογής. Είναι μια συγκεκριμένη, ένας συγκεκριμένος τρόπος, μια συγκεκριμένη απλούστευση αυτή. Υπάρχουν και άλλοι τομείς στους οποίους θα μπορούσαμε να αναφερθούμε, αλλά αυτό είναι κάτι ε, που μπορούμε να δείξουμε ότι έχουν καταβληθεί σοβαρές προσπάθειες. Τώρα, για την επιλεξιμότητα. Θέλω να θέσω αυτό το θέμα του ΦΠΑ. Ε, ένας από τους στόχους μας ήταν να υπάρχει κοινό κανόνας για τον ΦΠΑ. Ε, σε, υπό κάποια έννοια είναι αυστηρότερος από τον ισχύοντα, αλλά δεν νομίζω ότι προκαλεί σοβαρότερες δαπάνες, ε, δεδομένου ότι ο στόχος μας είναι ε, να εξασφαλίσουμε ότι όταν υπάρχει χρηματοδότηση ενός έργου υποδομής μέσω των δημοσίων οικονομικών, είναι δημόσιο ε, το έργο δηλαδή υποδομής, τότε ε, η χρηματοδότηση του ΦΠΑ θα, θα καταβάλλεται ο ΦΠΑ, ο οποίος θα πηγαίνει στον εθνικό προπολογισμό. Είναι λοιπόν θέμα εσωτερικών δημοσιονομικών ρυθμίσεων για το τι θα γίνει αυτός ο ΦΠΑ. Η, η άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι ότι δεν μιλάμε για δαπάνη αυτή καθεαυτή που πρέπει να χρηματοδοτηθεί από τον κοινοτικό προπολογισμό και ότι εφόσον μας ενδιαφέρει η βέλτιστη δυνατή χρήση των πόρων του προπολογισμού, ε, δεν πρέπει να προχωρήσουμε με αυτόν τον τρόπο. Ως προς τις κατηγορίες περιφερειών, η λογική που μας διέπει έχει επεξηγηθεί από την Επιτροπή και νομίζω ότι θα πρέπει να δούμε πώς έχει η πρόταση της Επιτροπής στο σύνολό της για το MFF ως προς το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Και θα πρέπει να δούμε πώς ορίζεται η δημοσιονομική μας πολιτική και πώς θα πρέπει να ενταχθεί ανάλογα με την πολιτική συνοχής και την Ευρώπη 2020 έτσι ώστε να έχουμε μία καλύτερη κλιμάκωση έτσι ώστε οι χρηματοδοτούμενες περιφέρειες να αντικατοπτρίζουν την πορεία προς μία πραγματική περιφερειακή ανάπτυξη. Θα πρέπει λοιπόν όλα αυτά να τα δούμε μέσα στα πλαίσια ενός συνολικού ισορροπημένου πακέτου. Δεν σημαίνει ότι εάν δεν υπάρχει αυτός ο συνεκτικός χαρακτήρας θα πρέπει η περιφέρεια να κινηθεί προς άλλη κατεύθυνση. Δηλαδή θα πρέπει να δούμε κατά πόσο αυτή η, κα κατηγοριοποίηση ε, συνάδει με τη δυνατότητα απορρόφησης. Ως προς τη μακροαιρεσιμότητα και τη συλλογιστική που μας διέπει, θα πρέπει να διατυπώσουμε τις ερωτήσεις ε, σωστά. Και το πρώτο είναι να δούμε κατά πόσο είναι λογικό να υπάρχει μια διαδικασία που να επιτρέπει την προσαρμογή της χρηματοδότησης για μια πολιτική συνοχής έτσι ώστε να υποστηρίζει τα εθνικά μέτρα για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τα υπερβολικά ελλείμματα ή τις μακροοικονομικές ανισότητες. Και η απάντηση είναι θετική. Θα πρέπει να υπάρχουν μηχανισμοί που να καθιστούν δυνατή την επανακατανομή πόρων για την πολιτική συνοχής για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε μια σοβαρή κατάσταση σε μακροοικονομικό επίπεδο. Γι' αυτό υπάρχει και ο μηχανισμός. Το δεύτερο ζήτημα είναι κατά πόσο είναι σωστό ένα κράτος μέλος το οποίο δεν έχει συμμορφωθεί με τις αποφάσεις του Συμβουλίου και τις συστάσεις του Συμβουλίου ως προς τα διορθωτικά μέτρα για να αντιμετωπίσει ένα υπερβολικό έλλειμμα ή μακροοικονομική ανισότητα θα πρέπει να λαμβάνει τις ίδιες επιστροφές από το, τον προϋπολογισμό για την πολιτική συνοχής ανεξάρτητα από την αποτελεσματικότητα αυτών των ε, μέτρων ακριβώς επειδή δεν πέτυχε να συμμορφωθεί. Η απάντηση είναι αρνητική. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε σαν να μην έτρεχε τίποτα. Κάτι συνέβη υπό τις συγκεκριμένες συνθήκες και θα πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι τα ευρωπαϊκά κονδύλια δεν εισραίουν προς ένα κράτος μέλος υπό μη βέλτιστες συνθήκες. Παράλληλα όμως θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρχει ευελιξία για την αναστολή πληρωμών. γιατί δεν μπορούμε να ξέρουμε εκ των προτέρων τις συνθήκες. Γι' αυτό υπάρχει ένα περιθώριο διακριτικής ευχέρειας, έτσι ώστε οι εισρωές να συνεχιστούν στα προγράμματα τα οποία θα πρέπει να τύχουν επένδυσης και η αναστολή να αφορά τα προγράμματα όπου δεν πρέπει να δοθεί συνέχεια. Επίσης θα πρέπει να επιδοτούμε ένα κράτος το οποίο βρίσκεται σε δυσκολίες εξαιτίας της μακροοικονομικής ε, κατάστασης και που την χάνει αρρωγής τη στιγμή που υπάρχει συμμόρφωση. Η απάντηση είναι καταφατική και γι' αυτό έχουμε αυτή την προσέγγιση top-up όπως ίσχυσε στην περίοδο μέχρι τώρα για να γίνει επιπρόσθετη χρηματοδότηση. Δηλαδή πρόκειται για μια συνεκτική προσέγγιση μέσα στα, στα πλαίσια αυτού του πακέτου μηχανισμών που είναι απόλυτα λογική. Τέλος, ως προς το Connecting Europe Facility, ε, ακούσαμε τους ε, συναδέλφους που είναι υπεύθυνοι για τον κανονισμό αυτό και τη διάδραση μεταξύ του ΣΕΦ και της πολιτικής συνοχής. Θα πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι λειτουργεί αποτελεσματικά γιατί θεωρούμε ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να γνωρίζουν μέσα στα πλαίσια της εξέλιξης των προγραμμάτων τους ποια προγράμματα μπορούν να τύχουν χρηματοδότησης με βάση το ΣΕΦ το Connecting Europe Facility. Γι' αυτό θεωρούμε ότι θα πρέπει να υπάρχει σαφήνεια ως προς τις προτεραιότητες για να υπάρχει μια σχετική προβλεψιμότητα από τα κράτη-μέλη για να μπορέσουν να προγραμματίσουν το μέλλον τους. Εάν το επιτύχουμε αυτό, τότε θα έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, δηλαδή θα έχουμε αυτά τα σημεία συνδέσμου των προγραμμάτων υποδομών, έτσι ώστε να χρηματοδοτούνται τη σωστή χρονική στιγμή για να μπορέσουν να συμβαδίζουν με τις δράσεις δυνάμει της πολιτικής συνοχής. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, Κωνσταντσα Κρέλ. Ευχαριστώ, Ντανούτα. Ίσως να προσπαθήσουμε να διευκρινίσουμε το εξής. Ο Λάμπερ και εγώ επιλέξαμε με τα λόγου γνώσεως τέσσερα σημεία από το έγγραφο εργασίας για να τα συζητήσουμε σε βάθος. Δεν έχει νόημα κάθε φορά το δύο ώρο που έχουμε στη διάθεσή μας να συζητούμε επί παντός του πιστητού. Αλλιώς δεν θα συζητούμε για τίποτα απολύτως. Γι' αυτό σας παρακαλώ να συγκεντρωθούμε σε αυτά τα θέματα. Γι' αυτό δεν θα πω τίποτα τώρα για τη μακροαιρεσιμότητα ή για το μέσο διασύνδεσης της Ευρώπης, Connecting Europe. Δεν είναι του παρόντος αυτό. Ε, στις επόμενες συνεδριάσεις της Επιτροπής θα τα συζητήσουμε εκτενέστερα. Να πω όμως μερικά απαντώντας εκείνους που αναφέρθηκαν στις τέσσερις σημερινές προτεραιότητες. Με χαρά. Ο συνάδελφος Γκοντμάνης ρώτησε ε, και τι μορφή θα λάβει η ευελιξία. Όταν κάποιος δεν κάνει κάτι καλά μπορεί να αλλάξει, να πάει σε άλλη προτεραιότητα. Ε, όχι, ακριβώς αυτό δεν θα είναι δυνατόν. Η ευελιξία θα συζητηθεί στην αρχή στη διαπραγμάτευση για τις συμβάσεις εταιρικέ σχέσει μεταξύ των τοπικών αρχών, των περιφερειακών, των κρατικών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στην αρχή θα ρυθμίζονται αυτά τα ζητήματα και θα πρέπει να κοιτούμε προσεκτικά να είναι σαφέστερη η διατύπωση για τον τρόπο με τον οποίο θα συμμετέχουν οι περιφέρειες, οι δήμοι και οι κοινότητες στην εκπόνηση αυτών των εταιρικών ε, συμβάσεων. Να το συζητήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να διευκρινίσει, να αποσαφηνίσει τι ακριβώς εννοεί και τι δεν εννοεί. Αλλά οι προθέσεις μας προς τα εκεί στρέφονται. Ελίζαμπετ Σρέντερ, άμα θες να το συζητήσουμε πολύ περισσότερο, ξέρω πολύ καλά ότι η δική μου πολιτική ομάδα στις τελευταίες διαπραγματεύσεις ήταν επίσης κατά του earmarking, ε, αλλά δεν είχαμε καμία ευκαιρία και το επέβαλε το κοινοβούλιο. Αν δούμε αναδρομικά τώρα τι συνέβη, η στρατηγική της Λισαβόνας απέτυχε. Και αυτή η προσημείωση στον προπολογισμό, το earmarking, είχε φτιαχτεί για τη διαδικασία της ε, Λισαβόνας. Από αυτό και μόνο όμως δεν βγαίνει τίποτα. Δεν επιτυχάνει κανείς τίποτα. Θα πρέπει να ξανασκεφτούμε και στις σημερινές προτάσεις για την ε, υλοποίηση των στόχων θα πρέπει να δούμε ποια είναι αυτά που εξυπηρετούν, τι είναι βοήθεια και τι είναι στενός κορσές για τις περιφέρειες, τις πόλεις και τους δήμους και τις κοινότητες. Οπωσδήποτε να τους αναγκάσουμε να εφαρμόσουν κάτι που δεν βοηθάει για τη μακροπρόθεσμη ε, ανάπτυξη. Και επίσης, ας το συζητήσουμε αυτό με τη δημοκρατική εξέλιξη. Βεβαίω και δεν είναι στόχος, αλλά είναι γεγονός και πρόκληση και κατά την άποψή μου, η αντιμετώπιση αυτής της πρόκλησης δεν γίνεται σωστά ε, με τα όσα λέει ο σημερινός κανονισμός. Θα δούμε πώς θα το διατυπώσουμε, πώς θα το οργανώσουμε, αλλά πραγματικά καλύπτεται πολύ λίγο για το τι θέλουμε στο μέλλον της πολιτικής συνοχής δεδομένης της δημογραφικής εξέλιξης. Και ο Γιάννη έκανε μια πολύ σημαντική ερώτηση, Όρμπριχτ. Πότε θα αποφασίσουμε για το περιεχόμενο, όταν θα έχουν κλειδώσει τα οικονομικά ή νωρίτερα. Έχεις απόλυτος δίκιο, Γιάν. Και ο Λάμπερτ και εγώ είμαστε πεπισμένοι ότι σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να αποφασίσουμε οριστικά δεν ξέρουμε τι προπολογισμό θα έχουμε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάνει προτάσεις πιο συντηρητικές από το Κοινοβούλιο. Και δεν έχουμε όσα κονδύλια είχαμε στη διάθεσή μας ε, την παρούσα προγραμματική περίοδο, αλλά λιγότερα. Και τι σημαίνει αυτό. Περικοπές. Θέλει το Συμβούλιο. Όταν κάνει περικοπές στο Συμβούλιο μπαίνει στην ουσία ε, της διαρθρωτικής πολιτικής και της πολιτικής συνοχής και θα πρέπει να το ξανασκεφτούμε. Τι μπορούμε ως πολιτική συνοχής να κάνουμε και τι δεν μπορούμε. Ελπίζω να έχει τη σοφία το Συμβούλιο να δεχτεί τις προτάσεις μας για να μην τα αναθεωρήσει, αλλά δεν το θεωρώ καθόλου απίθανο να μην χρειαστεί, ε, ε, να χρειαστεί να ξανασυζητήσουμε μάλλον. Χωρίς προπολογισμό δεν μπορεί κανείς να αποφασίσει για αυτά τα θέματα του ε, περιεχομένου και της ουσίας. Σε όλα τα υπόλοιπα θέματα που έχουν να κάνουν με τα τέσσερα σημεία που μας απασχολούν σήμερα, συμφωνούμε σχετικά, έτσι δεν είναι. Ξέρουμε τι θέλουμε, αλλά τώρα θα πρέπει να βρούμε μια ευφυή διατύπωση για να βοηθήσει και πολιτικά στην εφαρμογή και να μπει και με ένα σωστό νομικό τρόπο ως κείμενο του κανονισμού και να έχουμε και μια ισορροπία ανάμεσα στο γενικό κανονισμό και τους κανονισμούς τους επιμέρους για τα ταμεία, γιατί είναι πάρα πολύ στενή η σύνδεση. Ε, ε, ασχολήθηκα λίγο πιο εντατικά με την ανάπτυξη των πόλεων, θα τα συζητήσουμε και το Γενάρη. Είναι παντού, στο κοινωνικό ταμείο, στο ταμείο συνοχής, ε, στο ΦΕΝΤΕΡ, στο Γενικό Κανονισμό, στη Διασυνοριακή Συνεργασία και πάει λέγοντας. Θα πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ για να καταλάβουμε τι θέλουμε να πετύχουμε από κοινού και τι να εφαρμόσουμε. Και μια τελευταία παρατήρηση. Δεν αναφέρθηκα καθόλου στις ποσοστώσεις και ούτε κατά διάνοια συγκεκριμένα. Μάρτιν, δεν πιστεύω ότι είναι τόσο ευέλικτες οι περιφέρειες όσο δηλώνουν. Ας πούμε, στη Βόρεια Ιταλία, μια πιο ανεπτυγμένη περιφέρεια. Εκεί υπάρχει υποχρέωση. 52% του κοινωνικού ταμείου. Υπόλοιπο 48%. Από αυτό το 48% θα πρέπει να πάνε 5% τουλάχιστον για την αστική ανάπτυξη, υπόλοιπο 43% από το 43 80% για τις προτεραιότητες κλειδιά και το υπόλοιπο 20% ε, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αποδοτικότητα και μετά τι μένει. Γύρω στο 20% και με αυτό το 20% μπορώ να αρχίσω να κοιτάω τις υπόλοιπες προτεραιότητες ανάλογα με τις ανάγκες της περιφέρειας τελικά δεν είναι πολύ μεγάλο το περιθώριο λιγμών στις περιφέρειες και καμία ορατότητα ή προβολή. Λοιπόν, θα πρέπει να διαφυλάσσεται αυτή η ισορροπία, να κοιτάξουμε και να εξετάσουμε και να ελέγξουμε αν αυτό χρειαζόμαστε και θέλουμε πραγματικά. Γιατί δεν κάνουμε μια πολιτική συνοχής μόνο για το 2020, αλλά και για μια μακροχρόνια ανάπτυξη των περιφερειών που είναι και υποχρέωσή μας από τις συνθήκες. Αξίζει λοιπόν τον κόπο να το ξανακοιτάξουμε και να εξετάσουμε αν αυτή την ε, ευελιξία θέλουμε και χρειαζόμαστε στις περιφέρειες για να καυτούν και να καταργηθούν οι διαφορές και να έχουμε και αηφορονάπτυξη ταυτόχρονα. Ευχαριστώ. Ο κύριος Βανίσερόη ε, προεδρεύει Ευχαριστώ. Κυρία Χιούπνερ χρειάστηκε να βγει για λίγο, θα επανέλθει μάλλον και μου ζήτησε να προεδρεύσω εγώ. Ε, με χαρά, ευχαριστώ. Κυρία Κρέλ. Να προσθέσω κι εγώ μερικά πράγματα για την προσέγγιση. Και την άλλη φορά τέσσερις προτεραιότητες θα συζητήσουμε από το σύνολο, τα είπε ωραία η και ε, ίσως και αυτό που έχει να κάνει με τις σχέσεις των ταμείων ε, μεταξύ τους και τις θεματικές προτεραιότητες και τον κανονισμό. Να δούμε πώς πηγαίνει όλη αυτή η διακλάδωση των στόχων, αυτό το δέντρο των στόχων από την κορυφή μέχρι τη βάση. Να δω, όταν ψάχνω ας πούμε στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, και ψάχνω την ενέργεια ε, από πάνω μέχρι κάτω, δεν τη βρίσκω πουθενά. Μπορεί να φταίω εγώ και να πρέπει να ψάξω σε άλλο ταμείο. Αλλά μπορούμε να κάνουμε αυτή τη δουλειά στην άτυπη ομάδα εργασία Και προτείνω να είναι ξεχωριστό σημείο 9, 8, 10, 11, δεν ξέρω, δεν έχει σημασία, αλλά να το συζητήσουμε ε, γιατί έχει σημασία για τη λήψη των αποφάσεων. Πάντως ε, είναι πολύ μεγάλη προτεραιότητα για μας θα πρέπει να το συζητήσουμε και με τους άλλους συζητητές από τις ε, αντίστοιχες επιτροπές. Αυτά προς στιγμή στις τέσσερις επόμενες προτεραιότητες, κάπινγκ και λοιπά, η οροφή, ε, δεν θα τα συζητήσουμε τώρα. Προς το παρόν να τα αφήσουμε εδώ, να ευχαριστήσω όλους όσους μίλησαν και θα επανέλθουμε. Και τώρα το επόμενο θέμα είναι το σημείο 8 λέει εδώ. Εξέλιξη των μακροπεριφερειακών στρατηγικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τρέχουσα πρακτική και μελλοντικές προοπτικές, ιδιαίτερα στην περιοχή της Μεσογείου. Ο Φρανσουά Αλφονσί είναι εισηγητής μας για το θέμα αυτό. Έχετε το λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ανισχώ λίγο διότι ο σκιώδης εισηγητής που ήταν παρόν καθ' τη διάρκεια του απογεύματος, οι σκιώδης μάλλον, αποχώρησαν. Εκτός από ένα, αυτό το θέμα έπρεπε να συζητηθεί αύριο, μία ώρα. Τώρα μας μένουν 20 λεπτά. Αξίζει τον κόπο. Δεν θα ήταν ευγενικό και απέναντι στους σκιώδης που σηκώθηκαν και έφυγαν. Ήταν εδώ όλο το απόγευμα και τώρα έχουν φύγει. Δύο. Ο κύριος Ντόιτς και κάποιος άλλος. Υπάρχει κι άλλο θέμα πριν από μας ε, σήμερα το απόγευμα. Τα αεροδρόμια. Καλά, απουσιάζει ο εισηγητή η έκθεση πεπραγμένων της επίσκεψης αντιπροσωπεία στη Βαρσοβία. Δεν μπορούμε να συζητήσουμε αυτό και να ε, ακολουθήσουμε την ημερήσια διάταξη. Το θέμα προβλέπεται και αύριο το πρωί στι 9. δεν ξέρω, με λέγω μπερδεμένος, δεν ξέρω αν χειρίζομαι και τα μικρόφωνα. Έχετε δίκιο ότι είχε προβλεφθεί αρχικά για αύριο το πρωί. Έχετε απόλυτος δίκιο. Και πρέπει να συζητηθεί παρουσία των σκιωδών. Αλλά δεν μπορούμε να υποσχεθούμε ότι θα συζητηθεί μία ώρα ολόκληρη. Το θέμα ε, δεν είναι ε, η διάρκεια της συνεδρίασης αλλά η ουσία του θέματος και αν έχετε να πάρετε και αεροπλάνο γιατί είστε ειδικό για τα περιφερειακά αεροδρόμια πρέπει να το συζητήσουμε. Αύριο το πρωί μισή ώρα σας φτάνει, συμφωνείτε. Άντε, 40 λεπτά βαριά βαριά, μου λέει η γραμματεία. Εντάξει είμαστε, ωραία. Ε, συμφωνώ όλοι ο κύριος Αλφονσή Do you want to have it now? Ναι, ναι, συμφωνώ κύριε Πρόεδρε, προτιμώ. Ωραία. Και τώρα μας έχει απομείνει η έκθεση σχετικά με την επίσκεψη της αντιπροσωπείας της Επιτροπής μας στη Βαρσοβία, 16-17 Οκτωβρίου. Ποιος θα το πει. Έχουμε τα πρακτικά στη διάθεσή μας. Ήμασταν από την αρχή της Προεδρίας εκεί um, και μας ε, έκανε τον απολογισμό της Προεδρίας σήμερα η ε, Υπουργός. Συζητήσαμε αρκετά νωρίς, δεν ξέρω, κοιτώντας γύρω μου, ε, κοιτώ τους συναδέλφους αν θέλουν να κάνουν σχόλια. Μπορεί κάποιος να κάνει μία ανακοίνωση, να απλώ να ανακοινώσουμε ότι υπάρχει έκθεση πεπραγμένων και αν συμφωνείτε όλοι με τα πρακτικά είμαστε εντάξει. Δεν χρειάζεται να παρουσιαστεί και προφορικός. Κατά τη διάρκεια του εξαμήνου ε, επισκεφθήκαμε τη χώρα που προεδρεύει και νομίζω είναι καλό να συνεχιστεί αυτή η πρακτική. Έχουμε από πρώτο χέρι ενημέρωση στα αρχικά στάδια της προεδρίας. Ένα συνάδελφο ζήτησε το λόγο, κύριο Σόμπριχτ. Ε, ε, ήθελα να σας πω ότι κατά την επίσκεψη στη ε, Βαρσοβία επισκεφθήκαμε το Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και πολλά και σοβαρά ελέγχθησαν σε σχέση με τους νέους κανονισμούς και τα προβλήματα και τις δυσχέρες που υπάρχουν και γι' αυτό θα πρέπει οι εισηγητές ε, να μας υπενθυμίσουν τα σχόλια ενός κράτους μέλους κατά την Προεδρία αυτή. Ήταν πολύ σημαντική η συνάντηση με αυτά αποτελέσματα, άρα όταν συζητήσουμε τον κανονισμό ίσως θα πρέπει να τα υπενθυμίσουμε όλα αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ καλή αυτή η συμπληρώση, εξαιρετική. Και τώρα κοιτώ την ημερήσια διάταξη και διαπιστώνω ότι τελειώσαμε. Ολοκληρώνεται εδώ η σημερινή συνεδρίαση. Ραντεβού αύριο το πρωί στις 9 ε, για την υπόλοιπη ημερήσια διάταξη όπως έχουμε συμφωνήσει. Ευχαριστώ πολύ.